Παρακαλώ καθίστε. Υπάρχουν θέσεις πίσω. Ας μην επαναλάβω αυτά που είπα στην αρχή. Δηλαδή ας τα επαναλάβω. Ο, ιδέ, ο δεύτερος γύρος ομιλητών έχει εγκατασταθεί και τώρα θα ακούσουμε έξι επιχειρήσεις που ανήκουν σε πολύ διαφορετικούς τομείς, τις οποίες ευχαριστώ για την προσέλευσή τους, για να απαντήσουν στα ερωτήματα των συναδέλφων. Φίλιπ Μόρις, ΙΚΕΑ, Coca-Cola, Walt Disney, McDonald's και Anheuser Busch Inberg. InBev. Όπως κάναμε και για το προηγούμενο πάνελ, θα δώσουμε το λόγο στον κάθε εκπρόσωπο για να κάνει μία παρουσίαση το πολύ πεντάλεπτη και μετά θα ακούσουμε ερωτήσεις. Ίσως και απαντήσεις. Καταρχήν ο κύριος Βέρνερ Σούστερ, Vice President Tax του Philip Morris International. Μάλιστα, πρόεδρε μέλη, προσδοκώ στην ανταλλαγή απόψεων, αλλά προηγουμένως είπα λοιπόν, να σας κάνω λίγο το ιστορικό της Philip Morris International που είναι μια αμερικανική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη και στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Μας ανήκουν έξι από τις 15 μεγαλύτερες μάρκες τσιγάρων, ιδιαίτερα το Marlboro. Έχουμε πάρα πολλούς ε, εργαζόμενους που μιλούν 80 γλώσσες και λειτουργούμε 50 εργοστάσια στην Ευρώπη 12.000 εργαζόμενους και με εργοστάσια σχεδόν σε κάθε χώρα μέλος. Πέρυσι ανακοινώσαμε επενδύσεις 500 εκατομμυρίων για προϊόντα που μπορούν να μειώσουν τον υγειονομικό ατομικό κίνδυνο. Την τελευταία φορά που μετρήσαμε τα κέρδη μας έφταναν σε κάτι πάνω από 20 δισεκατομμύρια και είναι γνωστό ο φόρος που πληρώσαμε. 29,1% φόρο εισοδήματος πληρώσαμε. Και αυτά σας τα έχουμε στείλει. Τώρα πάλι για τους φόρους. Η προσέγγιση μας για τη φορολόγηση είναι η εξής συμμορφωνόμαστε με τους τοπικούς κανόνες. Οι αποφάσεις επιχείρησης δεν καθορίζονται από τα φορολογικά, είναι χωριστό. Πρώτα τα εμπορικά. Πληρώνουμε τους φόρους ανάλογα με τις δραστηριότητες μας σε κάθε χώρα. Είμαστε διαφανείς με τις φορολογικές αρχές στις χώρες όπου εργαζόμαστε, όπου λειτουργούμε δεν προσπαθούμε να αποφύγουμε ούτε έχουμε ιδιαίτερους φορολογικές δομές ούτε λειτουργούμε τις λεγόμενες letterbox companies. Συμφωνούμε ότι δεν έχουν συμμορφωθεί οι κανόνες της φορολόγησης με την παγκοσμιοποίηση και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα. Όποτε λοιπόν γίνεται ζητούμε περισσότερες εξηγήσει από τις φορολογικές αρχές της κάθε χώρας. Ε, να έχουμε μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα και αυτές και για μας. Τα tax rollings δεν είναι ο μόνος τρόπος. Στην Ιταλία ας πούμε θα συμμετάσχουμε στο συγκριτικό πρόγραμμα συμμόρφωσης μαζί με τις Ιταλικές φορολογικές αρχές και σε ανάλογο πρόγραμμα συμμετέχουμε και στην Αυστραλία. Αυτά είναι παραδείγματα διαφάνειας. Πολλές από τις ανησυχίες σας αφορούν ακριβώς το βαθμό διαφάνειας στα φορολογικά. Αυτά τα θέματα μόνο σε κυβερνητικό επίπεδο μπορούν να λυθούν. Και εμείς θεωρούμε τα εξής. Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες BEPS του ΟΣΑ, αλλά ανησυχούμε για την πιθανή άνηση εφαρμογή τους και με πιθανό αποτέλεσμα διπλή φορολόγηση. Ο μηχανισμός επίλυσης διαμαχών πολλές φορές έχει καταλήξει διπλή φορολόγηση. Η το κοινή φορολογική βάση που προτείνεται για την Ένωση θα μπορούσε να είναι κάτι αποδεκτό Συμφωνούμε επίσης για την αυτόματη συμμόρφωση με τα tax rules και δεν έχουμε αντίρρηση στις προτάσεις του ΩΣΑ για τις αναχώρασεις στάσης του. Για το βασικό μου θέμα της ε, διαφάνειας συμφωνούμε στις περισσότερες προτάσεις που κάνετε και εσείς και ο ΩΣΑ. Τα βρολικά καθεστώτα πρέπει να είναι διαφανή μεταξύ του φορολογούμενου και των φορολογικών αρχών και εμείς θα προσθέταμε και μεταξύ φορολογικών αρχών. Αν έχετε απορίες να μας τις λυπείτε. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Σημειώνω ιδιαίτερος μεταξύ των όσων είπατε ότι ο μιλός σας θα ήταν υπέρ όχι μόνο τη ενιαία φορολογική βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση CCTB για τη φορολόγηση των εταιριών, αλλά ακόμα και για ενιαίο συντελεστή θα συμφωνούσατε σε όλη την επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ερωτήσει και σχόλια μεταξύ των μελών μα. Ωραία. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο τη IKEA. Έπρεπε να το είχα πει από την αρχή. Ε, η σειρά με την οποία δίνεται ο λόγος είναι ανάλογα με τις απαντήσεις, τη χρονολογική σειρά ε, των απαντήσεων που έστειλαν οι εταιρείε. Πρώτη απάντησε η Google, γι' αυτό πήρε πρώτη το λόγο στο πρώτο πάνελ, έτσι είναι με χρονολογική σειρά. Και με αυτή τη σειρά δίνω το λόγο στον Κρίσον Μάτσον, τον αρμόδιο επικεφαλή των οικονομικών ε, θεμάτων στην IKEA. Έχετε το λόγο. Ε, Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ που με προσκαλέσατε και εμένα και την εταιρεία μου. Πριν σα πω την άποψή μου για το πρόγραμμα δράση ε, για το BEPS και την κοινή φορολογική βάση, να σα πω μερικά πράγματα για τον όμιλο IKEA. Στον κόσμο λειτουργούμε σε 40 αγορέ. Απασχολούμε 147.000 εργαζομένους παγκοσμίω και σε ό,τι αφορά τους φόρους πληρώνουμε 800 εκατομμύρια ευρώ σε εταιρικό φόρο με ένα φορολογικό συντελεστή λίγο κάτω από το 20%. Ο συνολικός λογαριασμός για τους φόρους με όλα τα, με όλα τα ποσά συμπεριλαμβανόμενα είναι περίπου 1,5 δις ευρώ. 31% των εισοδημάτων μας πριν φορολογηθούν αφορολόγητα δηλαδή τα καθαρά, τα ανοιχτά κέρδη. Έχουμε δικαιώματα να λειτουργούμε σε 28 χώρες και franchise ε, αυτές και επίσης 12 άλλες ομάδες με τέτοιες άδειες εκμισθωσής σε άλλες 22 αγορές. Η εταιρεία, η μητρική εταιρεία και το μεγαλύτερο μέρος του management βρίσκονται στην Ολλανδία. Δεν έχουμε κάποια θηγατρική στο Λουξεμβούργο. Ε, μας ελέγχει πλήρως το Ολλανδικό σύστημα και υπακούμε στην Ολλανδική φορολογική νομοθεσία. μπορούμε μόνο να επενδύσουμε τα προλικά έσοδα στον όμιλο. Λίγα λόγια τώρα για το σύστημα των Είναι ε, το σύστημα του franchise, ήταν κάτι που ξεκίνησε το 1980 η λιανική πώληση ε, διαχωρίστηκε από την ιδιοκτησία, τη μάρκα του, της IKEA και αυτό επέτρεψε και την επιτυχία του συστήματος franchise. Κάποιες φορές μας μπερδεύουν με τον όμιλο IKEA που είναι ξεχωριστός όμιλος. Όμως η βασική, το βασικό σύστημα δικαιοχρησιών και η μάρκα βρίσκονται στις κάτω χώρε είναι μέρος της μητρικής εταιρεία, ενώ ε, υπάρχει ξεχωριστός όμιλος στο Λουξεμβούργο, δηλαδή η εταιρεία μας αποτελείται από δύο διαφορετικά τμήματα. Να πω ότι ούτε ο ιδρυτής της εταιρείας, ο αρχικός ούτε ιδρυτής της εταιρείας, ούτε μέλη της οικογένειάς του έχουν τίτλους ιδιοκτησίας στον ε, έναν από τους δύο ομίλους, ό,τι αφορά το παγκόσμιο φορολογικό σύστημα να τονίσω την ανάγκη να υπάρξει εναρμόνιση του φορολογικού συστήματος που να είναι σταθερή και σαφής. Γι' αυτό το πρόγραμμα δράσης BEPS και γι' αυτό θελήσαμε και να έχουμε και ανταλλαγή απόψεων μαζί σα για αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα. Η επιτυχία του BEPS εξαρτάται από διάφορου παράγοντε, να φέρω μερικού. Πρώτα απ' όλα, είναι σημαντικό να υπάρχει συγχρονισμένη και συνεκτική υλοποίηση των συστάσεων σε ένα ε, σαφές εθνικό φορολογικό πλαίσιο. Ε, επίσης πρέπει να, υπάρξουν, να υπάρξει εφαρμογή των ρητρών για διατησία ε, δεσμευτικά για να αποφύγουμε φαινόμενα όπως η διπλή φορολόγηση. Κατά τρίτον, η υλοποίηση των συστάσεων BEPS πρέπει να είναι αποτελεσματική για να αποφευθεί το, το διοικητικό Τέλος, η Ευρώπη είναι μια από τις σημαντικότερες αγορές για τον ομίλο IKEA. 77% των εσόδων μας προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 47.000 εργαζομένους εδώ και 60% των προϊόντων μας ε, στην Ευρώπη. Θέλουμε να ε, προωθήσουμε περισσότερο την ε, παρουσία μας στην Ευρώπη και γι' αυτό η διαφάνεια και η σαφήνεια στο πολιτικό σύστημα μακροπρόθεσμα είναι ένα σημαντικός παράγοντας για μια εταιρεία σαν τη δική μας που θέλει να βρει επενδυτικές ευκαιρίες. ορίζουμε, λοιπόν κάθε προσπάθεια να βρεθεί μια κοινή λύση και σας ευχαριστώ πολύ για, τις λεπτομέρειες, για την φροντίδα στις λεπτομέρειες που δώσατε στη δουλειά σας. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία και αναμένω τις ερωτήσεις σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα θα πάρει ο κύριος Ρόμπερτ Φόρδον, αντιπρόεδρο του General Tax Council της Coca-Cola. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, για τα μέλη σας, εξ ονόματος της εταιρείας, που ξέρετε ότι εδρεύει στην Ατλάντα της πολιτείας Γεωργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, να σας δώσω κάποια στοιχεία για την εταιρεία μας και το δίκτυο εμφιάλωσης. Η εφεύρεση της Coca-Cola έγινε το 1886 στην Ατλάντα της Γεωργίας και μέχρι σήμερα εκεί ευρεύει ακόμα η εταιρεία. Είμαστε παγκόσμια εταιρεία, πολυεθνική, αλλά εργαζόμαστε σε τοπικό επίπεδο, ε, επιτόπου, στις τοπικές κοινωνίες. Από όλα τα ποτά μας που πουλούμε στον κόσμο, 81% πουλούνται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Αρχίσαμε τη λειτουργία μας στην Ευρώπη, στη Γαλλία το 1919. Σήμερα με τους εμφιαλωτές μας παράγουμε πάνω από 650 προϊόντα εδώ στην Ευρώπη σε 84 εργοστάσια σε 24 κράτη-μέλη. Με 48.000 άμεσα ε, απασχολούμενους και υποστηρίζουμε και 600.000 στην αλυσίδα διανομής, ε, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, εδώ και ένα αιώνα περίπου επενδύουμε στην ανάπτυξη, στην τοπική κοινωνία παντού στην Ευρώπη. Το σύστημα της Coca-Cola ε, συμπεριλαμβάνει την εταιρεία μας αλλά και πάνω από 250 εταιρείες εμφιάλωσης παγκοσμίω και έτσι έχουμε παγκόσμια κάλυψη με τοπική εστίαση. Δεν είναι από πλευράς διαχείρισης η νομικής ενιαία. Ε, οι περισσότεροι εμφιαλωτές μας είναι ανεξάρτητες εταιρείες. Ε, επίσης και ε, είναι φορολογούμενοι νομοταγείς σε όλες τις χώρες που λειτουργούν. Πληρώνουμε πολλούς φόρους στις χώρες αυτές, συμπεριλαμβανομένων ε, ειδικών φόρων ε, διαφόρων φόρων ε, κίνητης περιουσίας και φόρων για τα έσοδά μας. Το 2014 το λέει αυτό ο ισολογισμός μας και περίπου 2,2 δισεκατομμύρια αμερικάνικα δολάρια πληρώσαμε παγκοσμίω σε εταιρικό φόρο. Και ε, συντελεστής 23,6% σύμφωνα με το μέσο όρο του ΩΣΑ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που μας στείλετε και με χαρά να μοιραστούμε μαζί σας ε, τις πληροφορίες. Ε, σε ό,τι αφορά την ε, πρότασή σας για τα BEPS ε, του ΩΣΑ και τον εταιρικό φόρο ξέρω ότι ε, είστε υπέρ της ε, CCTV ενός, μιας ενιαίας βάσης για τη φορολόγηση. Εμείς είμαστε επικοδομητικοί στην προσέγγιση μας για το BEPS της πρωτοβουλίας του ΩΣΑ. Εάν εφαρμοστεί με τρόπο ενιαίο και υποκράτος δικαίου μπορεί να επαναφέρει την απαραίτητη εμπιστοσύνη στην φορολόγηση των πολυεθνικών ως πολυεθνική και παγκόσμια εταιρεία που το προϊόν προϊόντα σε 200 και πλέον χώρες, καλωσορίζουμε κάθε προσπάθεια για να βελτιωθεί η αξιοπιστία και να μειωθεί η περιπλοκότητα στη φορολογική συμμόρφωση. Θα πρέπει να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες που να εξηγούν ποιες ε, δραστηριότητες παράγουν αξία, κέρδος, για να συμφωνήσουμε όλοι πόσο ε, θα πρέπει να είναι εκείνο το ποσό των εσόδων ε, των εταιριών που επιχειρούν, που αναλαμβάνουν κίνδυνο. Εκτός από τα μέτρα BEPS που είναι η διάβρωση της βάσης και η μεταφορά των κερδών, θα πρέπει να δούμε και άλλε συστάσει του ΩΣΑ και να τι παρακολουθούμε ω προ την εφαρμογή του. Έτσι μόνο θα υπάρχει συνεκτική προσέγγιση και θα συμφωνήσουν και οι κυβερνήσει για να φορολογείται η εταιρεία στην ε, κατάλληλη χώρα κάθε φορά. Πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση, Αλλιώ. όταν υπάρχει τρομερή ε, αμφισημία ε, υπάρχουν πολλά περιθώρια για φορολογικέ αρχέ, για φορολογουμένους, υπάρχουν διαφορέ μεταξύ φορολογουμένων και κρατών και μεταξύ κρατών των ιδίων μεταξύ του, δηλαδή. Χρειάζονται συστήματα ε, υποχρεωτικής επίλυσης διαφορών για να λύνεται γρήγορα αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά την ενιαία βάση φορολόγηση εταιριών θέλουμε να μειωθεί η γραφειοκρατία, να αυξηθεί η προβλεψιμότητα και η ασφάλεια. Για να εφαρμοστεί αυτό το CCCTV θα πρέπει να συνεργαστούν οι κυβερνήσεις για να εναρμονίσουν ε, τους φόρους. Ε, αυτό βέβαια το εγχείρημα είναι τεράστιο και τρομακτικό και παραμένουν και άλλες προκλήσεις και άλλοι παράγοντε που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την επιχείρηση και τον κλάδο κάθε φορά. Το λέει και η εκθεσή σα. Το BEPS και το CCCTB είναι φιλόδοξοι στόχοι και για να επιτύχουν θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, υποστήριξη, αξιοπιστία μεταξύ τη εφορία των κρατών και των ε, πολιτών Για το φορολογουμένο Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσετε να συμμετέχουμε σε αυτή τη σημαντική συζήτηση. Και εγώ σα ευχαριστώ. Τώρα, ο Τζον Στάουελ από τον Walt Disney, Senior Vice President Corporate Tax. Πρόεδρε εξοχότατη, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Χαιρετίζουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις εδώ για τη γενική φορολογική πολιτική και ιδιαίτερα για το πρωτοβουλία BEPS του ΩΣΑ καθώς και την πρόσφατη πρόταση για μια κοινή φορολογική βάση στην συζήτηση. Εμείς καταλαβαίνουμε τη σημασία που έχει μια στεναρή φορολογική πολιτική και διαχείριση. Οι προοπτικές για τις επενδύσεις και η ανάπτυξη διεθνώς ενισχύονται όποτε οι φορολογούμενοι έχουν καλύτερη κατανόηση των φορολογικών κανόνων. Αυτό συμπεριλαμβάνει θέματα όπως το κατά πόσον οι δραστηριότητες μιας οντότητας πρέπει να φορολογηθούν ή όχι, καθώς και το πώς χρησιμοποιούνται τα κέρδη από την φορολογήσιμη αυτή παρουσία. Έτσι οι κυβερνήσεις μπορεί να λύσουν πιθανές φορολογικές διαφορές με ειρηνικό τρόπο. Επίσης υποστηρίζουμε τη συνεργασία με κυβερνήσεις για την απλοποίηση της διασύνδεσης των διαφόρων φορολογικών συστημάτων και γι' αυτό μας ενθαρρύνουν οι πρωτοβουλίες του ΣΑ και τα ΜΠΕΠΣ καθώς και από εσά ο υπολογισμός με απλούστερο τρόπο του, της κοινή φορολογικής βάσης επιχειρησιακής φορολογικής βάσης. Θα έπρεπε να προσθέσω ότι δεν αναμένω να υπάρξει καμία φοβερή διαφορά στη φορολόγηση από τον Πέψη το CCCTB διότι τα δικά μας κέρδη συμμορφώνονται απολύτως με τις οικονομικές μας δραστηριότητες και επειδή έχουμε πολλές δραστηριότητες σε χώρες με υψηλή φορολόγηση πληρώνουμε και παβολούς φόρους. Ως πολυεθνική με έδρα της Ηνωμένε Πολιτείε υποκείμεθα σε ποσοστό 35% αλλά το οποίο γίνεται 37% ή 38% μετά και από τους τοπικούς φόρους. Αυτό αναγνωρίζεται σαν από τις υψηλότερες φορολογίες στον κόσμο. Εκτός αυτού, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Φορολογικό Σύστημα, μας, όλα τα κέρδη φορολογούνται τελικά και στις Ηνωμένε Πολιτείες και καμιά φορά από τις ε, επιχειρήσεις στο εξωτερικό πρώτα πριν από τις τοπικές. Για το τελευταίο φορολογικό έτος, το Σεπτέμβριο φέτος, η εταιρεία μας ανέφερε 13,8 δισεκατομμύρια κέρδη με πάνω από 5 δισεκατομμύρια φόρους, δηλαδή 36% πραγματική φορολόγηση. Για τα τελευταία 4-5 χρόνια γύρω στα 34% είναι ο μέσος όρος φορολόγησης μας. Όπως θα περίμενε λοιπόν κανείς από μια εταιρεία τέτοιου μεγέθους, συν το μεγάλο φόρο εισοδήματος, ε, διακινούμε πάρα πολύ την τοπική οικονομία και γι' αυτό πληρώνουμε και συλλέγουμε και πολλούς έμεσους τόξους, τόκου, ε, φόρους. Συγχωρείτε. Επίσης, εκτιμούμε ιδιαίτερα μία θετική σχέση με τις κυβερνήσεις, με διαφάνεια, δικαιοσύνη, ακεραιότητα και εμπιστοσύνη. Όποτε είναι δυνατόν θέλουμε να λύνονται οποιασδήποτε διαφορές εκ των προτέρων ή διαφωνίες μεταξύ κυβερνήσεων ως προς το ποια χώρα πρέπει να φορολογήσει τη δραστηριότητά μας. Και ως αποτέλεσμα θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξουν μονομερείς ή διμερείς rulings αν αυτό καταλήγει σε μεγαλύτερη σαφήνεια για τις κυβερνήσεις ή τις επιχειρήσεις. Επίσης υποστηρίζουμε πρόσθετα μέτρα όπως incremental guidance για δραστηριότητες όπου κυριαρχεί κάποια ασάφεια ως προς τη φορολόγια εσύ. Υποστηρίζουμε την υποχρεωτική διαιτησία και οποιοδήποτε άλλο τρόπο επίλυσης διαφορών έτσι ώστε να υπάρχει ίση μεταχείριση και μεταξύ των φορολογουμένων. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την ευκαιρία και προσβλέπω και εγώ σε οποιασδήποτε απορίες θα θέλετε να σας λύσω. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Άιριν Γκέτς, που είναι αντιπρόεδρος των πολιτικών θεμάτων της McDonald's. Γεια σας, είμαι η Άιριν Γκέτς από την ομίλα McDonald's υπεύθυνη για τα φορολογικά θέματα, αντιπρόεδρος. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι ευχαριστώ να σας μιλήσουμε για, το, για τις προτάσεις για την κοινή φορολογική βάση και το BEPS του ΩΣΑ. Μερικές σύντομες πληροφορίες. Στην Ευρώπη βρισκόμαστε σε 39 χώρες, όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με περίπου 80.000 εστιατόρια εξυπηρετούμε 15 εκατομμύρια πελάτες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση παντού και απασχολούνται 350.000 εργαζομένους ενώ την Ευρώπη. 80% ε, των ε, πρώτων ε, των αγροτικών των τροφίμων που χρειαζόμαστε για την παραγωγή μας παράγονται στην Ευρώπη για την κατανάλωση της Ευρώπης. Τα τρία τέταρτα των εταιριών των εστιατορίων μας στην Ευρώπη τα έχουν αναλάβει εταιρείε δικαιοχρησία. Αυτό επιτρέπει να έχουμε μεγάλα κέρδη σε επίπεδο franchise. Και μακροπρόθεσμα έχουν άδεια να έχουν ένα σύστημα, ένα δικό τους εστιατόριο όσοι έχουν ε, τέτοια δικαιοχρησία και έναν ορίζοντα. Τώρα για την ε, φορολογία μας πληρώνουμε εταιρικούς φόρους σε όλη την Ευρώπη καθώς και κοινωνικούς φόρους, φόρους ακινήτων και επίσης το ίδιο και οι, όσοι έχουν, έχουν ε, δικαιοχρησία από εμάς franchise. Οι χώρες στι οποίε λειτουργούμε είναι οι χώρε βάσει των οποίων πληρώνουμε του φόρου. Από το 2010 στο 2014 οι εταιρείε McDonald's πλήρωσαν πάνω από 2,1 δι ε, δολάρια σε εταιρικού φόρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μέσο φορολογικό συντελεστή ήταν περίπου 27%. Ε, να σα δώσω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα από δύο διαφορετικέ χώρε. Στον Ηνωμένο μεταξύ 2009 και 2013, η εταιρεία μόνη τη πλήρωσε 2,9 εκατομμύρια ε, φόρους αγγλικές ε, ε, στερλίνες και στη Γαλλία την ίδια περίοδο πληρώσαμε πάνω από ένα δις ευρώ η McDonald's μαζί με, τις, με τα εστιατόρια δικαιοχρησίας και αναμένεται και για το επόμενο διάστημα να είναι πολύ ψηλά τα επίπεδα τη φορολογία μα. Τώρα, για το πώ πληρώνουμε του φόρου. Όπω τα συστήματα, τα συστήματα franchise συνήθω, οι ιδιοκτήτες μας, όσοι έχουν franchise ή και όσοι έρχονται κατευθείαν από τη μητρική εταιρεία, πληρώνουν ξεχωριστά, πληρώνουν ένα νητικό φόρο για την ε, χρήση του σήματος μεταφοράς και αυτό μας επιτρέπει να επενδύουμε περαιτέρω και να προχωρούμε σε καινοτομίε και εξελίξεις όλοι μας το σύστημα. Το όλο το σύστημα. Το σύστημα αυτό των royalties εξετάζεται πολύ προσεκτικά και το, και το ελέγχουν εξωτερικοί συνεργάτες με κρίσιμους δείκτες και μεθόδους του ΩΣΑ. Το ποσοστό που πληρώνεται είναι δίκαιο και βασίζεται στις ισχύουσες αρχές της αγοράς. Από την αρχή να ξεκαθαρίσω ότι ο τομέας αυτό είναι ιδιαίτερα περίπλοκος και γι' αυτό ίσω υπάρχει ατυχή μνήα της εταιρεία Μακτόλη στην Επιτροπή της, την έκθεση της Επιτροπή σα που λέει ότι έχουμε κερδοσκοπικέ μεθόδους φορολόγηση. Τώρα για τον ΟΣΑ, το BEPS και το CCTP ε, υπάρχουν κανόνες που ε, επηρεάζουν και τη λειτουργία, τη λειτουργία του δικού μας ομίλου. Στην φορολογία, ένα νέο σύνολο διεθνών κανόνων και κατευθυντήριων γραμμών θα επέτρεπε να έχουμε σαφέστερα, καθαρότερα, απλούστερα και συνεπέστερα φορολογικά συστήματα διεθνώ. Είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία ώστε οι πολυεθνικές να έχουν βεβαιότητα ως προς τις φορολογίε και θα θέλαμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πολιτικές συμφωνίες και στο μέλλον και δεν μας ε, δυσκολεύει καθόλου να παράσχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες αρκεί τις, εταιρείες, τις πληροφορίες για την εταιρεία μας να μην τις δημοσιοποιούν όσο τις λαμβάνουν. Ε, το σύστημα μπορεί να αναθεωρηθεί, αλλά δεν μας αρέσει η ιδέα της μονομερούς υιοθέτηση από χώρε και εφαρμογής, ε, διότι το σύστημα BEPS θα έπρεπε να εφαρμοστεί σφαιρικά και ταυτόχρονα. Ε, χρειάζεται συντονισμό για την επίλυση διαφορών από τι διάφορε χώρε και θα πρέπει να μην υπάρξουν εμπορικοί φραγμοί, ε, η προσέγγιση να είναι η άρση των φραγμών και όχι η δημιουργία νέων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει συνέπεια, νομική βεβαιότητα και σαφήνεια σε οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία σε αυτό το τομέα. Αυτό θα επιτρέψει την εταιρεία μα να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να πληρώνει τους φόρους εκεί όπου λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci, madame. Σας ευχαριστούμε. Και τέλος να δώσω το λόγο στον κύριο Μάλτε Λόχαν, στον όμιλο ΑΜΠΕ Président. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να έρθω αυτή τη σημαντική ε, σημερινή συνεδρίαση για να συζητήσουμε τα δύο αυτά θέματα που μας απασχολούν. Και θα συνεχίσω στα αγγλικά, μου επιτρέπετε. Λέγομαι Μάρτα ναι. Λόρν και είμαι αρμόδιος για τα παγκόσμια αυτά θέματα στην ΙΝΠΕΦ και τη θέση της για σημαντικά ε, θέματα πολιτικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς και μεταξύ αυτών φορολογικής πολιτικής η εταιρεία μας καλωσορίζει τις ε, συστάσεις της έκθεσής σας. Ε, πραγματικά θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω οι σημερινές συζητήσεις να συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση αυτή. Καταρχάς, να σας δώσω λίγο το υπόβαθρο για την InBev. Είμαστε παγκοσμίως πρώτοι στι ηθοποιίες και εδρεύουμε εδώ στη Λόβεν, έξω από τις Βρυξέλλες. Η Στέλλα Αρτουά και η Λέφε είναι σήματα γνωστά στο Βέλγιο, βαθιά ριζωμένα. Τελευταία, ε, τα τελευταία 700 χρόνια ορισμένε μπύρε. Ε, η Στέλλα Αρτουά μάλιστα ε, παράγεται στην ιστορική μας έδρα. 55 εκατομμύρια ευρώ θα επενδύσουμε έτσι ώστε να προωθήσουμε τη μάρκα Στέλλα παντού στον κόσμο. Να σας πω μερικά βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας. Ε, λειτουργούμε σε 25 χώρες και έχουμε πάνω από 155.000 εργαζομένους παγκοσμίως. Τα έσοδά μας το 2014 από αγορές από όλο τον κόσμο ε, είχαν ένα πλεόνασμα 43 δις ευρώ. Πληρώνουμε φόρους στις χώρες που λειτουργούμε. Το 2014 περίπου πληρώσαμε 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους παγκοσμίω και συμπεριλαμβανομένων 2,2 δις ευρώ σε φόρους εισοδήματος. Θα δείτε πολύ περισσότερες προφορίες στην ιστοσελίδα μας www.abpavlainbev.eu Τώρα για θέματα φορολογικά. Πρώτον, ε, το CCTV και μετά το BEPS. Υποστηρίζουμε ε, την έκκληση της Επιτροπής σας για ένα κοινό ενοποιημένο σύστημα βάσης φορολόγησης εταιριών. Θα πρέπει αυτό να βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές. Πρώτον, απλότητα. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα απλό, ε, χωρίς διοικητικά εμπόδια. Αυτό παραμένει σημαντικό εμπόδιο στην Ευρώπη. Συγγνώμη. Δεύτερον, ασφάλεια δικαίου για τις εταιρείε αλλά και για τις εφορίες. Τρίτον, σταθερότητα για να βοηθηθούν οι εταιρείε και να μπορούν να προγραμματίζουν μακροπρόθεσμα το σχεδιασμό του. Πιστεύουμε ότι η κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τι εταιρείε θα μπορούσε αυτά να τα εφαρμόσει στην Ευρώπη για να επενδύουν περισσότερο εταιρείε, να δημιουργούν θέσει εργασία και να προωθούν και να αναπτύσσουν την ευρωπαϊκή οικονομία καθώ και την ανταγωνιστικότητά τη. Η AB InBev καλωσορίζει αυτό που ζητάει η Επιτροπή σα για ένα μηχανισμό ε, ουσιαστικής και αποτελεσματικής επίλυσης των διαφορών ε, για τη διπλή φορολόγηση. Σήμερα η κατάσταση αυτή μπορεί να τραβάει και μέχρι 8 χρόνια και πολλά θέματα παραμένουν χωρίς επίλυση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι προτεραιότητα μια τέτοια ρύθμιση. Βεβαίως, ως εταιρεία ε, με παγκόσμια παρουσία χρειαζόμαστε φορολογικά συστήματα απλά και σταθερά παγκοσμίω, όχι μόνο στην Ένωση. Και εδώ έρχεται να παίξει σημαντικό ρόλο το σύστημα BEPS. Επειδή οι δράσεις επιτρέπουν ε, ευελιξία, θα πρέπει να εφαρμόζονται παντού με τρόπο συνεπή, παγκοσμίω, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τονίζουμε αυτό, έτσι ώστε να υπάρχουν ίσοι κανόνε παιχνιδιού ε, σε σχέση με την παγκόσμια οικονομία. Αυτό έχει να κάνει και με την ε, συνεχιζόμενη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Συνοψίζοντας, πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει η πολιτική φορολόγηση των εταιριών προς το καλύτερο, να υπάρχει ένα πλούστερο σύστημα με λιγότερα γραφειοκρατικά εμπόδια, περισσότερη ασφάλεια για εταιρείε και εφορίες και την απαραίτητη σταθερότητα για να εθαρρύνονται οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ελπίζουμε ο σημερινός μας διάλογος να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή και το στόχο και με χαρά ε, στην ανταλλαγή απόψεων να μπω και σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους για ένα πρώτο γύρο. Η πρώτη Εστέρ Ντελάνγκ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Παρακαλώ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Όπως και από τον προηγούμενο γύρο άκουσα τους ομιλητές να ζητάνε όλοι σαφήνεια από τους πολιτικούς και συνέπεια. Απευθύνομαι προς την εταιρεία Disney. Πρόσφατα δημιουργήσατε ένα ολόκληρο οικοδόμημα με 37 βήματα για να αφοφύγετε τη φορολόγηση. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν ο στόχος γιατί σίγουρα δεν ήταν ε, στόχος η σαφήνεια ούτε η διαφάνεια. Δεύτερον, μπορείτε να αρνηθείτε ότι στο Λουξεμβούργο τρεις θηγατρικές του Disney πλήρωσαν για τουλάχιστον έναν, τουλάχιστον μία πλήρωσε πολύ λιγότερο από ό,τι προβλεπόταν από την προηγούμενη περίοδο 9 με 13 αυτός ο υπάλληλό σας που σας το πέτυχε αυτό πρέπει να είναι ο πιο παραγωγικός από όλους. Έπειτα, άμα εφαρμόσουμε τους νέους κανόνες του ΟΣΑ είπατε δεν θα αλλάξουν πολύ οι φόροι σας γιατί σχετίζονται με την τοποθεσία. Έτσι ακριβώς είπατε. Πόσους κατοίκους έχει το Λουξεμβούργο, 550.000, άρα 2,8 δισεκατομμύρια κέρδη θα σήμαινε ότι ο κάθε Λουξεμβούργιος σας δίνει 5.000 ε, ευρώ κέρδη. Δεν νομίζω αν δω εδώ τους ε, Λουξεμβούργιους συναδέλφους ότι έχουν αντιδράσει. Παρακαλώ να μας εξηγήσετε λοιπόν αυτό τον αριθμό. Επίσης να σας διαβάσω κάτι από τα έργα που έχετε παραγάγει. Αυτά που γίνονται δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε και να γίνονται. Στα Σταχτοπούτα το έλεγε αυτό. Τέλος. Τα φορολογικά θέματα είναι μέρος του επιχειρησιακού σας προτύπου ή νομίζετε εκεί στο Disney ότι υπάρχει και μία ηθικολογική πλευρά. 0,8% φορολόγηση στο Λουξεμβούργο. Αν οι ουρές που γίνονται στην Disneyland του Παρισιού μετρήσετε πόσα κέρδη αποφέρουν. Είναι ηθικό να φορολογήσετε τόσο λίγο. Θέλω να μπορέσουμε να μάθουμε από αυτά όπως έλεγε και ο Lion King πάλι δικό σας έργο. Σας ευχαριστούμε στα χτωπούτα μας. Για τους σοσιαλιστάς ο Εμμανουέλ Μορέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ας αφήσουμε το Lion King γιατί θέλω να μιλήσω για το McDonald's τώρα. Ε, απασχολείται πολύ κόσμο στην Ευρώπη. Είπατε ότι πληρώνετε πολλούς φόρους. Θα ήθελα απλώς να σας θέσω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, την αλλαγή της δομής του ομίλου σας το 8 και το 9, δηλαδή η έδρα στη Γενέβη και η δημιουργία του McDonald's franchising στο Λουξεμβούργο για να πληρώνεστε και πνευματικά δικαιώματα από αυτό. Το 5,8% των luxemburgικών δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία αντιπροσωπεύεται. Αυτά όλα γίνονται για να βελτιστοποιήσετε τη φορολογία σας σε ολόκληρη την Ευρώπη και ειδικά στη χώρα μου. Μήπως προσπαθείτε να αποφύγετε τη φορολόγηση σε άλλες χώρες όπως την Ιταλία και τη Γαλλία και αν ναι, εγώ δεν βγάζω συμπεράσματα. Αυτές οι αλλαγές υπακούν αποκλειστικά στη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή διότι για το γαλλικό δίκαιο θα επρόκειτο για κατάχρηση. Δεύτερον, με τι μέσα παρά του 5,8% πνευματικά δικαιώματα το McDonald's franchising δεν πλήρωσε παρά μόνο 1,6% φοροεισοδήματο στο Λουξεμβούργο. Αυτού του αριθμού έχω. Και τέλος, για του μισθωτούς, διότι εμείς ενδιαφερόμαστε και για αυτούς τους σοσιαλιστέ. Η φορολόγησή σας αφορά και κάτι που μπορεί να ζημιώσει τους ε, μισθωτούς γιατί φαίνεται ότι σε μερικά εστιατόρια που έχουν άδειες franchises δηλαδή και που δεν λειτουργούν καλά έχετε φορολογική απαλλαγή. Πώς γίνεται αυτό. Αυτά είναι τα τρία ερωτήματα που ήθελα να θέσω στον εκπρόσωπο του ομίλου Μακδόναλτς. Για τους συντηρητικούς ο Μπέρντ Λούκε. Αντιπρόεδρος της ομάδας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω γερμανικά εγώ. Η ερώτησή μου απευθύνεται επίσης στην εκπρόσωπο της εταιρείας McDonald's. Σύμφωνα με ε, τα όσα διαβάζουμε στον τύπο, η McDonald's έχει 11 θηγατρικές σε φορολογικούς παραδείσους. Αλλά υπάρχουν παραπάνω ε, που δεν ε, κατονομάζει η εταιρεία McDonald's γιατί δεν οφείλει. Ισχύει αυτό λοιπόν για τις θηγατρικές που έχετε ως αριθμός σε χώρες που θεωρούνται φορολογική παράδειση. Είναι πολύ περισσότερες αυτές από 11. Γιατί κάτι ακούσαμε για τουλάχιστον 42 τέτοιες εταιρείες και καθόλου 11. Και πόσο ε, υψηλό είναι αυτός ο αριθμός των εταιρεών που έχετε εκεί των θηγατρικών σας. Που εμφανίζονται ε, να χρησιμοποιούν το όνομα με franchise. Ε, επίσης, μαθαίνουμε ότι εκείνοι που αγοράζουν, που νοικιάζουν ε, τη μάρκα σας, γιατί και συχνά πληρώνουν αυτά τα τέλη, σε μια δική σας θηγατρική στην ίδια χώρα, που ε, αυτό το 5% που κοστίζει το franchise το, το μεταφέρουν, το μεταβιβάζουν ε, σε μια άλλη θηγατρική σας σε φορολογικό παράδεισο. Ισχύουν όλα αυτά. υπάρχουν τέτοιες συναλλαγές με τα τέλη franchising και αυτές οι θηγατρικές σας ε, δεν παρέχουν υπηρεσίες εκείνους που χρησιμοποιούν τη φίρμα σας, απλώς την νοικιάζουν και παίρνουν τα λεφτά. Ευχαριστώ. Ο Νίλ Στόρβαλτς από τους Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μάλλον θα σας κάνω να βαρεθείτε, όπως μας κάνατε κι εσείς να βαριόμαστε. Θα μιλήσω για θέματα ηθικής και γούστου. Η ΚΕΑ θα ήταν καλύτερα να μας προσφέρει ένα γεύμα αντί να έρθει στο κοινοβούλιο. Σουηδικά και φτεδάκια με την ειδική του σάλτσα και την ε, σουηδική του ονομασία. Αυτά που λέτε ξανά και ξανά είναι ότι κάνατε το ίδιο που κάνουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή οι πολυεθνικές κάνουν όλες το ίδιο. Αυτή την απάντηση πήρα και από την ε, Μαρτίνα Ανκίτ όταν ε, είχε δοματίσει η απαγόρευση κυκλοφορία στα βράδια. Δεν, είναι, δεν νομίζω ότι είναι όριμος τρόπος να απαντάτε στις ερωτήσεις μας. Και γιατί. Γιατί οι φόροι χρησιμοποιούνται για τα δημόσια αγαθά Και αν δεν γνωρίζατε ότι υπάρχουν δημόσια αγαθά παλιότερα, θα μπορούσατε να το έχετε αντιληφθεί μεταξύ της βραδιάς της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου και του Σαββάτου 14. τα κάποια δημόσια αγαθά στο Παρίσι ε, έτυχαν μεγάλες κακομεταχειρίσεις Και για να σας πληροφορήσω σε εσά στη McDonald's ένας από τους αυτοσχέδιους βομβιστές ε, ουσιαστικά ε, ανατινάχθηκε μπροστά σε ένα τα δικά σα εστιατόρια. Άρα τα δημόσια αγαθά είναι απαραίτητα. Δεν μπορείτε να είσαστε ελεύθεροι σε αυτό το σύστημα. Κι όμως είσαστε αυτό ακριβώς. Αντίθεση καβαλάριδε. Τέρμα της ιστορίας. Ευχαριστώ πολύ. λοιπόν, θα δώσουμε τώρα το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Ο κύριος Σούστερ με την ίδια σειρά από τη Φίλιπ Μόρις. Ε, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι πολλές ερωτήσεις αφορούσαν τη Φίλιπ Μόρις. Μία μόνο. Εάν ε, ε, ασχολούμαστε με τα φορολογικά ναι, ασχολούμαστε, το λαμβάνουμε υπόψη, δεν είναι κάτι το οποίο ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις. Βεβαίως, όταν επενδύεις σε μια χώρα θες να επενδύεις σωστά και να κάνεις το σωστό, όχι μόνο από φορολογική σκοπιά, αλλά από εργασιακής, ε, φορολογικής, νομικής. Ε, μια επένδυση πρέπει να γίνει σωστά και ένα τμήμα αυτής της εξίσωσης είναι και οι φόροι. Αλλά δεν είναι το κίνητρο για εγκατάσταση κάπου. Δεν υπήρξαν άλλε ερωτήσει προς τη φίλη Μόρις. Κύριε ναι, ίσως να γνωρίζετε ότι το κάπνισμα προκαλεί πολλούς καρκίνους. Και είναι δημόσιο αγαθό η θεραπεία του καρκίνου και εσείς ε, αυτό το προκαλείτε και το αποφεύγετε. 29% περίπου φόρους πληρώνουμε ε, στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό σαν αναλογία. Ευχαριστώ κύριος Μάτσον από την ΙΚΕΑ. Ευχαριστώ επανέλθουμε στην πρόσκληση σε γεύμα. No, for it. Uh, what we... Δεν ε, το περίμενα αυτό. Αυτό που μας αρέσει πολύ σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται εδώ είναι ότι γίνεται πολύ ειλικρινής και ανοιχτή συζήτηση για να υπάρχει ένα μελλοντικό σύστημα σταθερό και διαφανές. Σε ό,τι αφορά ε, την αρχική πρόσκληση, είχαμε πει από την αρχή ότι εμείς δεν έχουμε ε, θυγατρικές ή μάλλον δεν έχουμε εκπροσώπους εδώ στην Επιτροπή σας και αν θέλετε να έρθουμε οι ίδιοι και όπως και ήρθαμε και χαρόμαστε πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Και σε σχέση με αυτό, καλέσαμε τα μέλη του Κοινοβουλίου να έρθουν μαζί μας ε, σε ένα γεύμα απλό. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό με πάσα ειλικρίνεια και πάσα ευσυνειδησία. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση για σας κύριε Μάτσον. Ε, ο κύριος ε, γιαν Χάιμερ, ε, με συγχωρείτε την προσπάθεια με βέβαιος, ε, μας έδωσε, μάλλον έδωσε μια συνέντευξη στην εφημερίδα Le Monde στις 30 Σεπτεμβρίου φέτος όπου δήλωσε ότι ο μιλός του δεν είχε καμία πρόθεση να αλλάξει τις πρακτικές φορολογικής βελτιστοποίησης, ε, με την επιφύλαξη βεβαίως ότι δεν θα αλλάξει και ο νόμος και ότι πλήρωνε κατά μέσο όρο 19% φόρο στο σύνολο των εισοδημάτων του. Νομίζω έτσι ε, μας είπατε κάτι για παραπάνω από 31%. Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε. Ναι, να το σχολιάσω. Είμαστε υπέρ των σχεδίων δράση Και αυτό είπα προηγουμένω για την καταβολή των φόρων. Είπα ότι έχουμε περίπου 21% ω ε, πραγματικό φορολογικό συντελεστή για του εταιρικού φόρου. Πληρώνουμε όμω επιπλέον και άλλου φόρου, επειδή και ιδιοκτησία έχουμε και πληρώνουμε και περιβαλλοντικού φόρου. Εάν τα προσθέσουμε όλα μαζί, ξεπερνάμε το 30% που σα είπα. Ε, φόρου που καταβάλλονται σε σχέση με το εισόδημα αφορολόγητο. Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η φόρη που εννοώ. Εάν προσθέσουμε και του τοπικού το ΦΠΑ, όλε οι εταιρείε πληρώνουν πάνω από 40% ε, σε όλε τι χώρε όπου, έχω, που δραστηριοποιούνται. Τέλος πάντων, ωραία, να δώσω το λόγο στον κύριο Τζόρντεν και να προσθέσω μια ερώτηση που και αυτή είναι ένα απόσπασμα από συνέντευξη ή μάλλον ένα παράθυμα, παράθεμα από έγγραφο των υπηρεσιών σας, της εταιρείας σας. Και επιβεβαιώνω αυτά που είπατε, σας καθησυχάζω. Στηρίζουμε τι φορολογικέ πολιτικέ που επιτρέπουν στι εταιρείε όπω η δική μα να λειτουργούν με ίσου κανόνε και σε ίσο ανταγωνισμό με τι εταιρείε εκτό Αμερική, των ΗΠΑ, που έχουν πολλά φορολογικά ωφέλη σε σχέση με τις επιχειρήσει που έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι αν μπορείτε κάπως να το ε, ε, εξηγήσετε. Τι φορολογικά ωφέλη εννοείται, ποια είναι αυτά τα ωφέλη που έχουν ε, επιλέξει εταιρείε οι οποίε δεν έχουν την έδρα στην Ατλάντα τη Γεωργία όπω εσεί. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Το σχόλιο για, το, για τους ισότιμους κανόνες και τις εταιρείε που έχουν την έδρα σε χώρες εκτός ΗΠΑ αναφέρονται κυρίω στο σύστημα το αμερικανικό για την ε, φορολόγηση διεθνώ. σε αντίθεση με την αναχώρα φορολόγηση τον κόσμο που έχουν συνήθω εδαφικό φορολογικό σύστημα ή σύστημα εξαιρέσεων έκπτωση από το φόρο. Για παράδειγμα, εμεί επενδύουμε ξανά στι χώρε όπου έχουμε δραστηριοποίηση και εφόσον φορολογηθούν τοπικά, αν τα χρήματα αυτά θέλουμε να τα ξαναφέρουμε στι ΗΠΑ ω εταιρεία που έχει την έδρα τη στι ΗΠΑ, θα πληρώσουμε έναν ε, φόρο προ αύξηση από αυτόν. Και ο φορολογικό συντελεστή στι ΗΠΑ είναι 35% από του πιο υψηλού στον βιομηχανοποιημένο κόσμο. Αν προσθέσετε και του ε, τοπικού φόρου, αυξάνεται ακόμη πιο πολύ. Οπότε, θα έπρεπε να πληρώσουμε φόρο προς αύξηση και για παράδειγμα, εάν είναι 25% ο φόρος μας σε μια άλλη χώρα, κάτι που συμβαδίζει περισσότερο με το μέσο όρο του ΣΑ, και τα ποσά τα ξαναφέρναμε στις ΗΠΑ σε 100 δολάρια εισοδήματος θα πληρώναμε 10 δολάρια παραπάνω φόρο στις ΗΠΑ. 10 δολάρια παραπάνω φόρο δηλαδή 65 μόνο από ε, τα 100 αυτά δολάρια εισοδήματο, θα μπορούσαμε να τα επενδύσουμε εκτός ΗΠΑ. Ενώ οι ανταγωνιστέ μα θα μπορούσαν να τα επενδύσουν απευθεία χωρί να πληρώσουν το φόρο προσάκτηση. Αυτό εννοούσαμε με του ισότιμου κανόνε και οι εταιρείε που έχουν την έδρα του στι ΗΠΑ ουσιαστικά ε, είναι σε δεσμενέστερη θέση σε σχέση με τι εταιρείε που έχουν έδρα αλλού στον κόσμο. Και για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, κάτι που σχολίασε κάποιο από του φιλελευθέρους, όπω συχνά έχει πει ο πρόεδρος του μήλου μα, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε το χρυσό τρίγωνο, δηλαδή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, κυβέρνηση και κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή μέσω αυτής της συνεργασίας θα μπορέσουμε να έχουμε και την άδεια και την κοινωνική αποδοχή για να λειτουργούμε στις χώρες όπου πουλάμε. Είναι σημαντικό λοιπόν το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και έχω πολλά παραδείγματα σχετικά να σας δώσω. Όπως την, ε, την πρωτοβουλία 5 προς 20 για χώρες της Αφρικής που ε, τους δίνεται ευκαιρία να ε, εργαστούν οι άνθρωποι εκεί, να στηρίξουν τις οικογένειές τους, να ενταχθούν στο εργατικό μας δυναμικό. Πιστεύουμε λοιπόν πολύ στην ανάγκη να στηρίζονται τα δημόσια αγαθά και τη στενή συνεργασία με, ανάγκη στενή συνεργασία με τι κυβερνήσει και την κοινωνία των πολιτών. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Τι θα απαντήσει στα χτωπούτα η Walt Disney. Ευχαριστώ. Το ερώτημα που τέθηκε βασίζεται σε παρεξήγηση. Υπήρξε μία αναδιάρθρωση όντως στην εταιρεία το 2009 για να απλοποιηθούν μερικές από τις δραστηριότητες μας εκτός ΕΠΑ και άρα να επαναχρησιμοποιήσουμε και να ανακατανύμουμε κεφάλαια. Το περισσότερο κέρδος που αναφέρθηκε ήταν, προέρχονταν από από πλήρως φορολογημένες δραστηριότητες. Άρα το να λέτε ότι ήταν πολύ χαμηλή η φορολόγησή του είναι παραπλανητικό. Γιατί είτε ήταν η holding company αυτή στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Αυστραλία ή αλλού, το ίδιο θα πλήρωνε γιατί είχαν ήδη πληρωθεί και φορολογηθεί, εισπραχθεί και φορολογηθεί τα κέρδη και αυτό σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανόνες. Γι' αυτό δεν είχαν υποβληθεί σε πρόσθετο φόρο εισοδήματος. για τις άλλες δραστηριότητες, οι είδη δραστηριοτήτων υπήρξε μια χρηματοδότηση που έγινε με μιας αμερικανικής, ενός αμερικανικού κλάδου μας και γι' αυτό οι ΙΠΑ είχαν το δικαίωμα να φορολογήσουν εκείνο το κέρδος και γι' αυτό προβλέψαμε να συμμορφώνονται πλήρως τα κέρδη μας με τις δραστηριότητες που όπου είχαν δημιουργηθεί. Για να σας πω τώρα. Εμείς χαιρόμαστε πολύ για την παρουσία μας σήμερα εδώ και θα ήθελα να επαναλάβω μερικά πράγματα. Συμφωνούμε πλήρως, συμμορφωνόμαστε πλήρως με τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους και ταυτόχρονα στηρίζουμε την μεγαλύτερη σαφήνεια και καθαρότητα ως προς τους συνολικούς μας φόρους. Είναι πολύπλοκο θέμα, αλλά θέμα όπου χρειάζεται μεγαλύτερη απλοποίηση και σαφήνεια και από την κυβερνητική πλευρά και από την πλευρά των επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση που αναφέρατε πριν, που πολύ λίγη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων μας έγινε μέσω Λουξεμβούργου και το ποσοστό που επιβλήθηκε τόκου ήταν σύμφωνο με τις ισχύουσες διαδικασίες και το tax ruling που έθεσαν οι αρμόδιες αρχές. Αν θεωρείτε ότι έπρεπε, θα έπρεπε στο μέλλον να ακολουθηθούν διαφορετικοί κανόνες, εμείς θα ήμασταν υπέρ της προώθησης του κοινού μας στόχους της μεγαλύτερης αφήνειας και απλότητας. Θα πρόσθετα δε ότι το μεγαλύτερο τμήμα των διπλωματικών μας δικαιωμάτων που εισπράττουμε και άρα φορολογούμεθα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μεγαλύτερο αυτό ποσοστό είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πληρώσαμε πάνω από 5 δισεκατομμύρια μόνο και μόνο για φόρους εισοδήματος τον τρέχοντα φορολογικό χρόνο. Άρα είμαστε υπέρ οποιονδήποτε μέτρων θα κατέληγαν σε δικαιότερη σε δικαιότερο φορολογικό σύστημα σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε και που θα διευκόλυνε και τα διαμεθοριακά καθώς και την αύξηση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν απαντάει. Το θέμα του κύριου στόχου της αναδιάρθρωσης που αφορά όπως σας είπα τουλάχιστον 34 διαφορετικά βήματα. Clarity. What was the primary... Αυτός ήταν ο κύριος στόχος. Και εγώ έχω τέσσερις ή πέντε διαφορετικές πηγές που επιβεβαιώνουν τους αριθμούς που σας ανέφερα. Ποιο τμήμα αρνείστε για την περίοδο 9 με 13 δημιουργήσατε ή όχι τρεις θηγατρικές στο Λουξεμβούργο και ένας μόνο υπάλληλο τις διοικούσε και τις τρεις και οι θηγατρικές αυτές αφορούσαν ή όχι 2,8 δισεκατομμύρια όχι 2,8 άμα δείτε το εισόδημα το οποίο αφορά το Λουξεμβούργο αυτό το εισόδημα εξαιρείται της φορολογίας. Όπως θα γινόταν και για τη Γαλλία, αν ήταν στη Γερμανία, στη Γαλλία και αλλού. Ως τον αριθμό των υπαλλήλων, οι περισσότεροι υπάλληλοι της χρηματοδοτικής οντότητας βρίσκονται στη ΣΥΠΑ και γι' αυτό εκεί φορολογήθηκαν και όχι στο Λουξεμβούργο διότι βάζουμε μαζί, αντιστοιχούμε τη δραστηριότητα με το κέρδος και τη φορολόγηση. Γι' αυτό ήταν τόσο μικρή η φορολόγηση στο Λουξεμβούργο. Και το θέμα του Ernst και Young με τα 34 βήματα. The reason why, um, uh, Κοιτάξτε, αυτό το σχέδιο ήταν για να έχουμε μία δομή holding company ώστε να μπορέσουμε να αναχρησιμοποιήσουμε τα κεφάλαιά μας στην Ευρώπη με κύριο όφελος το ότι όλες αυτές οι οντότητες είχαν ε, ιδιοκτησία Ηνωμένων Πολιτειών και θα έπρεπε να φορολογηθούν κατά 35%. Άρα χρησιμοποιώντας τη holding company μειώσαμε κάπως αυτόν τον παραπάνω αμερικανικό φόρο. Και ο λόγος που είναι τόσο πολύπλοκο με 34 βήματα είναι γιατί ήταν πολλές οι οντότητες που μεταφέρθηκαν και πολλές οι χώρες. Δεν είναι και τόσο ασυνήθιστο. Αλλά σχετικά απλός ο στόχος. Δεν είναι τρομερός ο αριθμός των βημάτων αυτό. Ευχαριστώ. Μακδόναλτ τώρα. Ε. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις ε, ε, απευθύνθηκαν σε μένα. Θα προσπαθήσω τώρα να απαντήσω. Πρώτον, σε ό,τι αφορά ε, τις ε, διαρθρωτικές αλλαγές στη Γενέβη και στο ε, δικαιοχρησία στο Λουξεμβούργο. Κοιτάξτε, αυτό είναι στοιχείο της επιτυχίας μας. Ε, έτσι δουλεύουμε με αυτό το σύστημα franchise. 73% των ε, εστιατορίων στην Ευρώπη, σχεδόν 3 τέταρτα εργάζονται και δουλεύουν αυτό το σύστημα franchise και πληρών loyalty στην, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη φύρμα και διάφορα άλλα στοιχεία και τις, τα πνευματικών δικαιωμάτων χρησιμοποιούν τη μάρκα McDonald's και δεν χρειάζεται ε, να ε, εφευρίσκουν οι ίδιοι κάποια στοιχεία από ε, το franchise. Τώρα, πώς δίνουμε εμείς τις άδειες και με ποια κριτήρια και ποιο είναι το σύστημα που λειτουργούμε παγκοσμίω. Τα τέλη καταβάλλονται και από δικά μας εστιατόρια, της ιδιοκτησίας δηλαδή και της δικαιοχρησίας. Και αυτό γίνεται ε, με βάση κάποιες κατευθύνες γραμμές του ΩΣΑ για να έχουμε ένα ποσοστό τέλους που θα πληρώνει ε, σε εκείνον που νοικιάζει τη φύρμα προς το McDonald's. Έχουν γίνει διαφορετικές αλλαγές, δικαιολογημένες και απολύτως στοιχειοθετημένες. Και στην Γαλλία και την Ιταλία είχαμε διάφορα προβλήματα και προκλήσεις τα τελευταία χρόνια. Αλλά το McDonald's, μια στιγμή να σας δώσω και τα ακριβή στοιχεία, και αυτά είναι δημόσια. Ε, το 2010 στο 2014 ανοίξαμε πάνω από χίλια νέα εστιατόρια στην Ευρώπη και δημιουργήσαμε 500 54.000 άμεσες θέσεις εργασίας, για να μην μιλήσω για τους προμηθευτές. Τα, ε, οι συντελεστές για τα τέλη, για το franchising, τα loyalty διαφέρουν από χώρα σε χώρα και ε, ίσως εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη εναρμόνιση στο μέλλον. Ειλικρινά δεν κατάλαβα το θέμα αυτό που ρωτήσατε για ε, τα πρόστιμα και τους μισθούς. Μακδόναλντ θεωρεί, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το ρόλο ε, της ως εργοδότη. 420.000 εργαζομένους έχουμε και τους δίνουμε και πριν. Και επίσης τους εκπαιδεύουμε <laughs> και ε, έχουν και άλλες παροχές. Ε, τώρα, για τις θηγατρικές. 11 είναι ο σωστός αριθμός Ας ρωτήστε. Κοιτάξτε, εμείς λειτουργούμε σε 119 χώρες. Και όπου δραστηριοποιούμαστε, είτε είναι δικά μας τα εστιατόρια, είτε είναι με franchise, και αυτοί κάποια εταιρεία θα στήσουν. Και αν υπάρχει McDonald's σε φορολογικό παράδεισο, καταρχήν σας συνιστώ να πάτε να φάτε εκεί. Και ε, δεν είμαι βεβαία ότι έχω τις προφορίες που με ρωτάτε. Thank you. How about the, excuse me, how about the past? Ο κύριος Λούκε. Ναι, αλλά τι γίνεται με αυτή τη μεταβίβαση των εσόδων, ε, των τελών που πληρώνει κάποιος για να νοικιάσει τη φίρμα για να πάρει το franchising αυτό και τα μεταφέρουν σε φορολογικούς παραδείσους. Πώς γίνεται αυτή η μεταβίβαση. Πληρώνουν royalties, είπαμε, στις εταιρείες που έχουν τις άδειες και τις νοικιάζουν είναι ένα συνδυασμός του συστήματος που ισχύει στι Ηνωμένε Πολιτείε για τι ανώνυμες εταιρείε εξαρτάται από χώρα σε χώρα. Όχι, συγγνώμη, λέει ο κύριο Λούκε. Μπορείτε να αποκλείσετε το ενδεχόμενο ότι οι πληρωμέ των τελών από κάποιον που έχει τη δικαιοχρησία και έχει νοικιάσει τη φύρμα από μια θηγατρική. Εσείς μπορείτε αποκλείεται το γεγονός ότι αυτά πάνε σε φορολογικούς παραδείσους. Εξαρτάται ποιος δίνει την άδεια, ποιος την νοικιάζει. Και ξέρετε η εταιρεία αυτή ε, ε, χρηματοδοτεί και ενοτομία, ανάπτυξη. Ναι, αλλά ε, αν πάει μέσα από τη θηγατρική που έχει την φύρμα και την νοικιάζει, γιατί να πληρώνει και δεύτερη. Καλά, Υπάρχει, υπάρχει τρόπος συλλογής, μπορείτε να μας δώσετε στοιχεία για τον αριθμό 42 που σας είπα και όχι 11, ναι θα επανέλθω με διευκρινήσεις, διότι το μοντέλο αυτό του franchise είναι σαφές ως επιχειρηματικό, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να παίρνει αυτά τα έσοδα ε, εάν δεν έχει λάβει την άδεια, δεν έχει νοικιάσει με σύμβαση ε, που συνδέεται αυτό και με κάποιους κινδύνους και ανάληψή τους. Και έτσι έχει το δικαίωμα κανείς να συλλέγει τα τέλη. Ωραία. Θα μας δώσετε αυτή την απάντηση γραπτός και τώρα ο κύριος Μορέλ θέλει να κάνει μια συμπληρωματική ερώτηση, διευκρινιστική. Μάλλον δεν με καταλάβατε για τους μισθούς αυτό που ρώτησα. Εγώ δεν μιλούσα για το επίπεδο μισθών του McDonald's, δηλαδή πόσο παίρνουν, παρόλο που ξέρουμε ότι είναι μικρά τα ποσά αυτά. Αλλά υπάρχουν ομοσπονδίες ευρωπαϊκών συνδικάτων που έχουν βγάλει λαγό. Μήπως ε, εμφανίζεται τεχνητές ζημίες στο franchising για να μην παίρνουν πριν οι εργαζόμενοι. Αυτή είναι η ερώτηση. Διαφωνώ ότι δημιουργούμε τεχνητά εμπόδια, τεχνητές ζημίες. Εμείς θέλουμε παντού να έχει κέρδη επιχείρησή μας και να αναπτύσσεται σε όλες τις χώρες που λειτουργεί. Ευχαριστώ. Ε, Άρα είναι η ανετική απάντηση. Ο κύριος Λόχαν, να προσθέσω απλώς μια ερώτηση για τους φίλους από την ΑΜΠΕ ΙΝΠΕΒ. διότι διαβάζοντας εφημερίδες Διάβασα στη New York Times στις 20 Οκτωβρίου τρέχοντος μία δήλωση Βέλγου Υπουργού που ερωτήθηκε από Αμερικανό δημοσιογράφο λέγοντας ότι το βελγικό σύστημα ε, έχει σχεδιαστεί για να ελκύει η θέση αναπασχόλησης και να υπάρχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα σε τομείς όπως η παραγωγή ποτών, υποτοπία, όπου ζηθοποιία όπου η χώρα αριστεύει εδώ και αιώνες. Εδώ θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το συγκεκριμένο αποτέλεσμα από το γεγονός ότι στο Βέλγιο εταιρείε όπως η δική σας υπολογίζοντας χονδρικά τα φορολογίσμα κέρδη στο Βέλγιο μπορεί να ωφεληθούν με ένα σύστημα που ονομάζεται νοητή ε, νοητό επιτόκιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα για τα ερωτήματα της κυρίας Δελάνγκη και του κυρίου Μορέλ. Και μετά θα πάω στη δική σας ερώτηση. Το φορολογικό σύστημα έχει να κάνει και με τις αποφάσεις που λαμβάνουμε για την επιχείρησή μας. Προφανώς το αν σε μερικές χώρες βρισκόμαστε μόνο για τα φορολογικά του συστήματα είναι όχι απάντηση και να εξηγήσω τι εννοώ. Η μπύρα είναι μια παραγωγή ιδιαίτερα τοπική. Έχει σχέση και με την πολιτιστική κληρονομιά που αναφέρατε. Βεβαίω κάποιε μάρκε τι πουλάμε, τις πουλάμε σε όλο τον κόσμο, σε πολλέ χώρε. Αλλά κυρίω έχουμε τοπική παρουσία. Με μάρκε διαφορετικέ από την ε, μια χώρα στην άλλη. Οπότε εξαρτώμεθα πολύ από την κατάσταση που επικρατεί στην κάθε αγορά. Προκειμένου να καθορίσουμε στη συνέχεια και τι αποφάσει μα για το πώ θα λειτουργήσουμε, τι επενδύσει μα και τη φορολογία. Αυτό αφορά και τι υποδομέ μα, τι εγκαταστάσει, το τι δεξιότητε θέλουμε να έχουν οι εργαζόμενοι μα. Βέβαια, ξέρετε και από την σταθερότητα ενό πολιτικού συστήματο σε κάθε χώρα, το πόσο εύκολα διασυνδέεται τη χώρα με τι άλλε και το κάθε εξή. Η φορολογία είναι φυσικά ένα από τα κριτήρια, αλλά δεν είναι πάντα ποτέ η κατευθυντήρια από το κατευθυντήριο στοιχείο. Οι φορολογικοί συντελεστέ είναι ένα σημαντικό παράγοντα, αλλά και άλλα στοιχεία των φορολογικών συστημάτων, όπω το κατά πόσο είμαστε βέβαιοι ότι οι κανόνε θα ισχύσουν, η σταθερότητα του φορολογικού συστήματο, η δυνατότητα επίλυση διαφορών. Είναι ορισμένα παραδείγματα, τα έχω αναφέρει και προηγουμένω. Οπότε, Αυτό που είπαμε και από την αρχή για τη διαδικασία BEPS και CCTV. Ε, σίγουρα θα μπορέσουμε να κάνουμε μια διαφορά, γιατί σίγουρα αυτό θα κάνει μια διαφορά στις αποφάσεις που θα λάβουμε για τι επενδύσεις μα και το κατά πόσον θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε σε αγορέ τη Ευρώπη ή εκτός. Τώρα για τι μειώσει των νοητών ε, επιτοκίων, των νοητών τόκων στο Βέλγιο. Αυτή είναι μια δυνατότητα που δίνεται σε κάθε εταιρεία στο Βέλγιο. Ισχύει για όλους, οπότε και για μας. Και η ιδέα πίσω από αυτό το σύστημα είναι κάτι που συζητιέται αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο επίπεδο της εταιρικής φορολογίας. Είναι μια μορφή εταιρικής φορολογίας και η συλλογιστική για αυτό το είδος την προσέγγιση είναι να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ε, τη ταξιόγραφα και όχι από τις μετοχές και όχι αυτές που χρηματοδοτούνται από τα χρέη. Οι εταιρείε δηλαδή κάνουν ε, περισσότερες επενδύσεις κατά αυτόν τον τρόπο και νομίζουμε ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα για το φορολογικό πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής και καλό να το σκεφτεί, όντως. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τώρα να περάσουμε στην δεύτερη στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Ο κύριο Βιέγκας, εξ ονόματο της Ενωμένη Αριστερά. Καλησπέρα, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Έχω μια πρώτη ερώτηση προς τους εκπροσώπους της IKEA και της McDonald's. Μπορεί βεβαίως να ισχύει και για τους υπόλοιπους και έχει περισσότερο να κάνει με το τι θα γίνει στο μέλλον. Ακούσαμε κάποια τυπικά παραδείγματα για επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και για μετατόπιση των κερδών σε χώρες όπου δεν φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο τα κέρδη. Δηλαδή, εταιρείε που έχουν τα εργοστάσια του σε μια συγκεκριμένη χώρα, ε, αξιοποιούν του πόρου τη χώρα αυτή, όμω μετά δεν συμβάλλουν στην ανανέωση των εγκαταστάσεων που έχουν στη χώρα αυτή, προσπαθούν τα κέρδη να τα πάνε αλλού για να υποφεληθούν από όλα αυτά που γνωρίζουμε. Και αυτό αντίθετα με τις διάφορες αξίες που ευαγγελίζονται, τις αξίες που λένε ότι υποστηρίζουν και το καθεξής. Και αυτό γίνεται σε επίπεδο ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων γεωγραφικών ζωνών όπου υπάρχουν αναπτυσσόμενες χώρες. Οι πρακτικές λοιπόν αυτές είναι γνωστές και πρέπει να δούμε κατά πόσον συμβάλλουν αυτές οι μεγάλες πολυεθνικές ε, ε, σε μια αλλαγή της νοοτροπίας. Τι μπορούν να κάνουν οι πολυεθνικές, οι μεγάλες πολυεθνικές και να κάνουν κάποια πράγματα διαφορετικά από ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Ένα συγκεκριμένο λοιπόν ερώτημα προς την Coca-Cola. Και έχει να κάνει με πολύ συγκεκριμένε μας ε, ε, ανησυχίες, αυτές των Ισπανών εργαζομένων. Η Coca-Cola Βεβαίω συμμετέχει σε αυτά τα συστήματα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Υπάρχουν από την άλλη και προσπάθειε αναδιάρθρωση ανακατανομές των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε όλη την Δυτική Ευρώπη. Το θέμα λοιπόν είναι ποιες χώρες θα πληγούν περισσότερο και τι θα γίνει με τα εργοστάσια της Ισπανίας. Ευχαριστώ. Η κυρία Εύα Ζολή, εξ των Πρασίνων, αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προς διευκόλυνση της επικοινωνίας θα ρωτήσω στα αγγλικά. Πρώτη ερώτηση προς την Κοκακόλα η ευρωπαϊκή αγορά είναι 10% περίπου ε, του παγκοσμίου τζίρου σας και δεν ξέρουμε ε, πόσους φόρους πληρώνετε στην Ευρώπη. Ξέρουμε όμως ότι η ελληνική εταιρεία εμφιάλωσης, η δεύτερη μεγαλύτερη, ε, που δημιουργήθηκε στην Αθήνα στη δεκαετία του 50, τον Απρίλιο του 2013, άλλαξε την έδρα της αποφάσισε να φύγει από την Αθήνα και να εγκατασταθεί ε, στο, ε, στην Ελβετία, στη Ζηρίχη και να είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Περιέργως, αφού ε, αυξήθηκε ο συντελεστής του εταιρικού φόρου στην Ελλάδα μετά από πιέσεις της Τρόικας. Και σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις, αυτό οδήγησε σε οικονομίες πάνω από 30 εκατομμύρια ε, για το 2013 ε, από φόρους που δεν καταβλήθηκαν στην Ελλάδα αλλά πήγαν στην Ελβετία. Ξέρουμε ότι είναι η κατάσταση δύσκολη και πάρα πολύ δρακόντια τα μέτρα λιτότητας και θέλω να σας ρωτήσω για ποιο λόγο η Coca-Cola ενέκρινε να φύγει 3 ε από την Ελλάδα και να πάει στην Ελβετία αν δεν ήταν να αποφύγει να πληρώσει εκατομμύρια φόρων στην Ελλάδα, όπου είναι η πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Και μια ερώτηση προς την IKEA. Προσπαθήσατε το 2009 να κάνετε φορολογική συμφωνία με το Λουξεμβούργο. Τι φόρους πληρώνετε σήμερα στο Λουξεμβούργο και τι γίνεται με τις θυγατριές σας στην Ολλανδ... Ε, στις Ολλανδικές Αντίλες, στην ε, Ελβετία και στην Κύπρο. Και ε, για τη Φίλιπ Μόρις, πάρα πολύ σύντομη ερώτηση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο έχετε πέντε θηγατρικές στην ίδια διεύθυνση στην Ολλανδία. Μαυρούν Μιλάν 20, Μπέργεν Οπζούμ. Σε αυτή τη διεύθυνση πέντε θηρίδες και στην Ελβετία υπάρχουν άλλες θηγατρικές ε, που πληρώνουν τα τέλη τους. Για ποιο λόγο, στην Ελβετία. Και μια τελευταία ερώτηση προς όλους. Θα θέλαμε να μάθουμε το κόστος των τελών που πληρώνεται για ε, φοροτεχνικούς και άλλους τέτοιου συμβούλους εσωτερικούς και εξωτερικούς. Αυτό ρώτησε και το πρώτο πάνελ, ρωτήθηκε και το ξαναρωτάτε και στο δεύτερο πάνελ. Η κυρία ε, Μπάρμπαρα Κάπελα από την ΙΕΝΕΦ e για δύο λεπτά. Α, ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη, δεν σας είδα. Ξέχασα το Μάρκο, αν είναι δυνατόν. Ξέχασα το Μάρκο ε, από την FTD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο συγκεκριμένε ερωτήσει για την McDonald's και την IKEA. Και μετά μια γενική για όλους. Για την McDonald's αμφισβητήσατε τους αριθμούς του Tax Justice. Ε, μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής που πληρώσατε στο Λουξεμβούργο το 2013. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό τουλάχιστον. Για την IKEA. Μπορείτε να μας πείτε λίγο καλύτερα, να μας εξηγήσετε τι έλεγχος υπάρχει στην Ευρώπη με τη δομή που έχετε, γιατί όπως μας είπατε, φαίνεται σαν να είσαστε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει την έντρα της στην Ολλανδία. Αλλά έχετε 35 δις ευρώ περιουσιακά. Δεν νομίζω λοιπόν ότι ο σκοπός σας είναι να μην, πραγμα... να μην υποφελείστε τα κέρδη. Ε, και μια ερώτηση που αφορά όλους τους εκπροσώπους των ομίλων, των εταιριών. Η κάθε εταιρεία στον Όμιλο, με τη διοργάνωση, τη διάθεση που μπορεί να έχει στην Ευρώπη. χρησιμοποιείτε τα ivory loans, τα υβριδικά δάνεια μεταξύ των ε, μετρικών και των θηγατρικών εταιριών και πώς φορολογούνται οι ε, χρηματικές ροές μεταξύ των ε, μετρικών εταιριών, των εταιριών holding και των θηγατρικών. Πώ είμαστε βέβαιοι ότι φορολογούνται έτσι που πρέπει. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Τώρα έχει το λόγο η Μπαρμπαρά Κάπελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Κάπελ από την ΕΝΕΦ. E Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή ε, των εκπροσώπων των εταιριών στη σημασία που αποδίδουμε εμεί, Μια μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας δείχνει ότι ετησίως τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάνονται μέχρι και 70 δισεκατομμύρια ευρώ από εταιρικού φόρους και μέχρι 190 δις ε, υπάρχουν ε, ε, διάφορες ρυθμίσεις είναι ένα τρίτο παραπάνω από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Είναι τεράστια τα ποσά αυτά και γι' αυτό το κοινοβούλιο μας έχει αντιδράσει όχι μόνο με τη σύσταση της έκτακτης επιτροπής αλλά και με άλλες εκθέσεις. Εμείς έχουμε μια έκθεση κατά της επιθετικής φορολογικής πολιτικής, αυτόματη ανταλλαγή ε, ε, πληροφοριών και ε, ενιαία βάση για φορολόγηση. Ακούω ότι συμφωνείτε και καλωσορίζετε να υπάρξει ένα CCTB ενιαίο για τις εταιρείες στην Ευρώπη. Εμείς ως Κοινοβούλιο στους φορολογικούς συντελεστές είμαστε ακόμα πιο ευέλικτη. Κάποιος από εσά είπε ότι ε, θα θέλατε και έναν ενιαίο συντελεστή. Ο ανταγωνισμός είναι σημαντικός στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι διέξετε θετικά υπέρ της πρωτοβουλίας BEPS ε, του ΩΣΑ και αυτό μας αφορά και μας το Κοινοβούλιο και το δίκαιο ανταγωνισμού. Και σας ερωτώ γιατί από ό,τι βλέπω υπάρχει συναντήληψη από όλες τις εταιρείες. Έχετε εταιρείε ή θηγατρικέ σε φορολογικού παραδείσου και αν ναι, όπω είπε το McDonald's, ε, εν ώψη των σημερινών εξελίξεων και αυτά που συζητούμε εμεί, τι θα κάνετε. Μήπως ε, εταιρείε που έχουν θηγατρικές σε φορολογικούς παραδείσους θα σταματήσουν να παίρνουν επιδοτήσεις από την Ένωση, θα σταματήσουν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ευρωπαϊκούς. Ε, τι θα κάνετε, ε, χρησιμοποιείτε θηρίδες και ναι, ε, πώς το δικαιολογείτε στη δημιουργία αξίας. Γίνεται λόγος για ένα σήμα δίκαιης φορολόγησης, fair tax label. Σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Θα σας ενδιαφέρει να έχετε ένα αριθμό φορολογικού μητρώου, ένα αφημί ευρωπαϊκό. Ε, και πώς θα αντιμετωπίζετε όλα αυτά τα θέματα. Ωραία. Και η, η φορολογική δήλωση αναχώρα επίσης. Απαντούν με την ίδια σειρά. Πρώτος ο κύριος Σούστερ. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συγκεκριμένη ερώτηση για τη φίλη Μόρις πέντε ε, εταιρείε στην Ολλανδία όπως είπατε μία στο, στην Ολλανδία όπως είπατε μία στο Ντόρμουν στο Άμστερνταμ Έχουμε εταιρείε σφραγίσματο στην ε, Ολλανδία και εργοστάσια για ε, ημιτελή προϊόντα και ε, παραγωγή και δύο εταιρείε holding στην Ολλανδία. Πέντε όλα αυτά. Εάν πληρώνουν φόρου στην Ελβετία. Μερικές από τις εταιρείες αυτές έχουν υπηρεσίες management από την Ελβετία διότι κάποιες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το κέντρο του management στην Ελβετία και πληρώνουν αμοιβέ management στην Ελβετία. Η δεύτερη ερώτηση ήταν για τις αμοιβέ για τους συμβούλους. Ε, δύσκολο να απαντήσω συγκεκριμένα στην ερώτηση, διότι προφανώς στον εταιρικό φόρο έχουμε και τις αμοιβέ των ε, συμβούλων μας, αλλά έχουμε και τόσες θηγατρικές στον κόσμο που ε, τους Ευρωπαίους συμβουλούς τους έχουμε σε τοπικό επίπεδο, αλλά πολλές φορές έχουμε πτώσει λόγω φόρων ειδικής κατανάλωσης, λόγω ΦΠΑ και ούτω καθεξής σε εταιρικό επίπεδο στο δικό μας φορολογικό πεδίο νομίζω το συνολικό ποσό ε, που καταβάλουμε στους συμβούλους μας είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Για τους υπόλοιπους, για τις υπόλοιπες δικατρικές θα μπορούσα να κάνω μια εκτίμηση, αλλά προτιμώ να μην την κάνω. Ε, Συνήθω πάντως έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίε για την ε, παρακολούθηση της συμμόρφωσης Τώρα για τους εταιρικούς φόρους, σίγουρα εταιρείε στον ομιλό μας χρειάζονται κάποιο ρευστό, ενώ κάποιες άλλες είναι πλούσιες σε ρευστό. Αυτό τι, ε, γίνεται, υπάρχει τόκος, λίμπορ, ε, περίπου 8% όταν υπάρχει δανεισμός από μία εταιρεία χωρίς ρευστό, από αυτήν που έχει ρευστό μάλλον σε αυτήν που δεν έχει. Τώρα η εταιρεία που δίνει το ρευστό θα μπορούσε να είναι στη Γαλλία, τη Γερμανία, όπου τύχει να βρίσκεται η εταιρεία που έχει ρευστό στα χέρια τη. Αλλά το περιθώριο είναι πολύ μικρό, 1,36% περίπου, γιατί η εταιρεία απλώς εντοπίζει το που βρίσκεται το ρευστό, που βρίσκονται τα μετρητά και από που μπορεί να τα πάρει. Ε, αυτοί λοιπόν που αναλαμβάνουν, σύμβουλοι που αναλαμβάνουν αυτό, ε, παίρνουν κάποια κέρδη παρόμοια με μια τράπεζα για τη δουλειά τους είναι ακριβώς αυτή. Γι' αυτό κάνουμε μελέτε συγκρισιμότητα για να είμαστε βέβαιοι ότι οι αμοιβέ που δίνονται στι εταιρείε που μεσολαβούν είναι σωστέ. Μια άλλη ερώτηση δόθηκε για τα 70 δι που χάθηκαν από το φρονικό εισόδημα λόγω μετατόπιση κερδών. Είναι δύσκολο να γνωρίζει κανεί το ακριβέ ποσό. Είναι 70, είναι 40 δι. Είναι μεγαλύτερο από 70 δι. Οι πρωτοβουλίε που συζητήθηκαν στην Επιτροπή σα νομίζω ότι θα βοηθήσουν να βεβαιωθούμε ότι το εισόδημα φορολογείται εκεί που υπάρχει και δραστηριοποίηση και εκεί που υπάρχει προστιθέμενη αξία. Η μετατόπιση των κερδών εάν βασίζεται σε εταιρείε φαντάσματα ή σε τέτοια διάρθρωση πλασματική δεν νομίζω ότι γίνεται αλλά είναι και δύσκολο να καταλάβει κανείς ποιο είναι το ακριβές ποσό για το φορολογικό ανταγωνισμό νομίζω πάντοτε κίνητρα θα αναζητά κανείς Εάν μια χώρα έχει χαμηλό φορολογικό συντέλεστη, ακόμη και με την κοινή φορολογική βάση, γι' αυτό το σχολίασα προηγουμένω, εάν ισχύει το σύστημα CCCTB, θα πρέπει να είναι ενιαίο ο φορολογικό συντελεστή, διότι αν υπάρχει αυτό, ε, θα πρέπει να υπάρξει και ευθυγράμμιση, μάλλον να υπάρχει φορολογική βάση του εισοδήματο ανά χώρα. Αλλά κάποιε χώρε φορολογούν ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων και το εισόδημα. Εάν λοιπόν κανείς έχει ένα εργοστάσιο που έχει πολλούς εργαζομένους, εάν δεν έχει το ίδιο φορολογικό συντελεστή σε όλη την Ευρώπη, ε, θα πάει στη χώρα που έχει το βολικότερο φορολογικό συντελεστή. Οπότε οι κλίδες κατανομής θα εξυπηρετούσαν την ε, εταιρεία που βρίσκεται στη χώρα με το χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή. Και τώρα με το σήμα τη δίκαιη φορολόγηση. Θα μπορούσαμε να το δεχτούμε και να είμαστε υπέρα, αλλά το θέμα είναι Ποιο θα το αποφασίζει αυτό το σήμα, ποιε θα είναι οι προαπαιτήσεις, οι προποθέσει. αν η δικασία θα είναι ανοιχτή και διαφανή. Αλλά εάν ισχύσει αντικειμενικά, ευχαριστώ θα τη στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ίσως η κυρία Ζολή θέλει να ρωτήσει κάτι ακόμα. Μπορείτε να μα στείλετε γραπτό το ακριβές ποσό του τι πληρώνετε στους συμβούλους σας για τα φορολογικά και οικονομικά θέματά σας. Ευχαριστούμε. Ο κ. Μάτσον. Για την ΙΚΕΑ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι ξανά. Γιατί ορισμένες από τις ερωτήσεις αφορούσαν το, ε, μια, ένα άλλο, μια θηγατρική εταιρεία της IKEA. Ο ιδρυτής της ΙΚΕΑ ήθελε να παραμείνει η IKEA ως έννοια και στο μέλλον. Και το έχει μεταβιβάσει λοιπόν αυτό και τη φίρμα σε ένα ίδρυμα. Και σε ό,τι αφορά τους φορολογικούς παραδείσους ή τα εξωτικά νησιά, εμείς δεν είμαστε εκεί πουθενά παρόντες και πληρώνουμε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ φόρους το χρόνο. Για να επανέλθω στην ερώτησή σας κυρία Ζολή, δεν έχουμε τέτοιες εταιρείες θηγατρικές. Αυτά ανήκουν στο ίντεκ και είναι άλλος όμιλος και δεν τα ξέρω καθόλου. Εξ όσο γνωρίζω αυτό που λέτε είναι ανακριβές. Διότι ο πρόεδρος του Ιντερ ε, Ινκέα λέγεται Ματίας Κάμπρα και δεν μπορεί να είναι συνωνυμία ή τυχαίο. Και ο Γιώνας Κάμπρα είναι ε, ε, ο πρόεδρος του Ίνκα Holding βέβαια, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία holding ο Ματίας και ο Γιώνας είναι και στο εποπτικό συμβούλιο μιας τρίτης εταιρείας που την, ε, την ε, ε, η ιδιοκτησία έχει η οικογένεια Κάμπραντ. Λοιπόν, μην μας λέτε ότι είναι δική σας εταιρεία, δική σας είναι και παρά είναι και δεν απαντήσατε και στα προηγούμενα που σας ρώτησα. Ναι, επανέρχομαι στο τελευταίο σχόλιο. Οι ιδρυτές έχουν μια εταιρεία που ονομάζεται Econ και είναι η ιδιωτική τους περιουσία, είναι σαφές αυτό. Σε ό,τι αφορά τον Ματίας Κάμπρατ, είναι στο εποπτικό συμβούλιο της IKEA και ο Γιώνας Κάμπρατ, ένας από τους γιους, είναι και επίσης μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου. Για μας είναι ξεχωριστό το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ο έλεγχος των εταιριών και δεν υπάρχει συνδιαχείριση, ούτε κοινό management. Και δεν ξέρω τι κάνει η IKEA και ο όμιλος αυτός. Αν θέλετε έχουν πάρα πολύ καλή ιστοσελίδα και μπορείτε να βρείτε από εκεί όλες τις προφορίες. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, δεν είμαστε παρόντες πουθενά σε εξωτικά νησιά και φορολογικούς παραδείσους υπό την έννοια αυτή. Και πληρώνουμε φόρους, ε, το Ίδρυμα Ίγκα, ε, ε, σύμφωνα με την νομοθεσία. Στην Ολλανδία επίσης Κάποιος είπε ότι δεν πληρώνουμε φόρους. Βεβαίως και πληρώνουμε. Έχουμε 3.000 εργαζομένους και πληρώνουμε 25% εταιρικό φόρο κανονικά και η εταιρεία διαχείρισης ε, λειτουργεί στο Λάιντεν της Ολλανδίας ε, και είναι η έδρα μας παγκόσμια. Είμαστε πάρα πολύ ενεργοί και δραστήριοι στην Ολλανδία όπου και πληρώνουμε όλους μας τους φόρους. Και επανέρχομαι τώρα ε, τι πληρώνουμε σε φοροτεχνικούς ε, για την ε, συμμόρφωση, γιατί είμαστε σε πάνω από 40 χώρες, είναι πολύ περίπλοκες οι νομοθεσίες και εκεί έχουμε συμβούλους και φοροτεχνικούς βεβαίως που τους πληρώνουμε για να μας ελέγχουν τη συμμόρφωσή μας. Σε ό,τι αφορά τις ενδομιλικές συναλλαγές και δανειοδότησεις χρησιμοποιούμε για πολύ μακροπρόθεσμες επενδύσει στις μετοχές. Α πούμε τώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε να εγκατασταθούμε στην Ινδία όπου χρηματοδοτούμε πλήρως ε, με μετοχές ε, όταν είναι τόσο μακράς πνοή η επένδυση και ε, χρηματοδοτούμε μία εταιρεία την άλλη ενδομιλικές συναλλαγές πάντα βασιζόμενοι στα επιτόκια της αγοράς και στα ισχύοντα με κάθε διαφάνεια και ε, ε, εκεί πέρα τηρούμε και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΩΣΑ. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις για την ΙΚΕΑ και ορισμένε από τις άλλες που κάνατε ε, δεν αφορούν το IKEA Group, είναι άλλοι, άλλοι όμιλοι και έγινε κάποια παρεξήγηση. Très bien. Je vous remercie. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα... Να πάμε στην Coca-Cola. Ο κύριος Τζόρνταν. <clears throat> Uh, Ευχαριστώ. Η πρώτη ερώτηση ήταν ε, για την Χελένη CCHPC, έναν από τους συμφελωτές μας και τη μετακίνηση από την Ελλάδα στην ε, Ελβετία. Η Coca-Cola Hellenic έχει καταγωγή ελληνική και έχει σημαντική παρουσία στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Όμως, η μετακίνηση από η μετακίνηση προς την Ελβετία είχε είχε σκοπό και, καλύτερα, και να ανέβει η έχει στο χρηματιστήριο και να έχει περισσότερη πρόσβαση στα κεφάλαια, στις χρηματαγορές και να ανεβάσει τα εισοδήματά της και τη δυνατότητα επενδύσεων. Παραμένει στην, η εταιρεία στην Ελλάδα, θα έχει 24 δις ευρώ επενδύσεις στην Ελλάδα σύντομα, οπότε παραμένει ελληνική ε, η παρουσία της εταιρείας αυτής και διατηρεί ε, τα εμφυλωτηριά της στην Ελλάδα. Ως προς τη δεύτερη ερώτηση για του Ευρωπαίου εταίρους, εταίρους της Coca-Cola, πρόσφατα ανακοινώθηκε μια ε, συναλλαγή, μια συγχώνευση καλύτερα, μιας ισπανικής μας εταιρείας, της Αϊμπηρία, με μια γερμανική που λειτουργεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λόγος για τη συγχώνευση αυτή είναι ότι κάθε μια από τις εταιρείες αυτές έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα ατού. Λόγος της συγχρονεύσης, λοιπόν είναι να συνδυαστούν αυτά. Δηλαδή το ισπανικό εμφιαλωτήριο έχει μεγάλη παρουσία στα μικρά καφέ, στα εστιατόρια γενικώ, ενώ ο Γερμανός εμφιαλωτής έχει μεγαλύτερους λογαριασμούς, μεγαλύτερους πελάτες και σε, μια δύσκολη, σε ένα δύσκολο οικονομικό τοπίο στην Γερμανία. Η CCB λοιπόν όπως λειτουργεί και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ειδική εμπειρογνωμοσύνη ως προς τη δυνατότητα να λειτουργεί να λειτουργεί σε πάνω από μία χώρες. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για την συγχώνευση και αυτό για να συνδυάσουμε βέλτιστες πρακτικές των δύο εταιριών και να έχουμε έναν ισχυρότερο ουσιαστικά εμφιαλωτή με παρουσία σε πολλές χώρες ανά την Ευρώπη. Τέθηκε και μια ερώτηση για το 10% του συνολικού μας κύκλου εργασιών, το οποίο το κερδίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστός ο αριθμός, βάσει της έκθεσης του 2014. Αυτό είναι ο κύκλο εργασιών, το ποσοστό των κύκλων εργασιών που έχουμε στην Ευρώπη τα περισσότερα χρόνια. Είναι σημαντικό να σκεφτούμε όταν κοιτάζουμε τον κύκλο εργασιών έναντι του κατεβληθέντος φόρου ότι αυτά εξαρτώνται και από τα περιθώρια της εταιρεία. τη επιχειρηματική δραστηριότητα, μάλλον. Αν υπάρξουν πολλέ δαπάνες σημαίνει ότι υπήρξε και πολλή δραστηριοποίηση. 100%. του κόστους των δαπανών μας, να συγκρίνουμε δηλαδή όχι απλώ τον κύκλο εργασιών, αλλά το φορολογήσιμο κέρδος ε, σύγκριση με τα ποσά που καταβλήθηκαν. Διότι αν δούμε μόνο το φόρο που έχει καταβληθεί, είναι κάπως παραπλανητικό αυτό. θα δείτε ότι οι φόροι, μας, οι που πληρώνουμε συμμορφούνται με τον μέσο φορολογικό συντελεστή σε όλο τον ΩΣΑ και στις εταιρείε φιάλωσης. Ε, επίσης για τη συμβουλευτική. Βεβαίω και έχουμε συμβουλευτική. 200 χώρε πουλάμε τα προϊόντα μα. Πολλέ έχουν πολύ περίπλοκα φορολογικά συστήματα. Οπότε έχουμε φοροτεχνικού και υποστήριξη για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε σε αυτό το δύσκολο σε αυτή τη δύσκολη θάλασσα της φορολογίας και κάποιες φορές έχουμε πολύ συγκεκριμένε διευθεντήσεις στην ε, συνεργασία με τους φοροτεχνικούς. Εξηγήθηκε και στο προηγούμενο πάνελ λέγοντας γιατί δεν συμφωνούμε με αυτές τις πρακτικές. Επίσης συμφωνούμε με το σύστημα CCCTB Επί της αρχής υπάρχουν δυσκολίες στην υλοποίηση, όπως η εναρμόνιση της βάσης ή ποιοι θα πρέπει να είναι οι παράγοντες που θα καθορίζουν, αλλά η Επιτροπή σας είπε ότι καλωσορίζει την έκθεσή μας. Ε, να έχουμε υπόψη ότι διάφορα θέματα επιμέρους μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθούν. Η τιμολόγηση λόγου χάρη και το τι γίνεται με τα κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με συγχωρείτε. Ναι, ναι, έχω μια συμπληρωματική ερώτηση. Η Coca-Cola πιστεύει ότι χρειάζεται η έδρα σας να βρίσκεται στο Ζουγ για να έχετε καταχώρηση στο Λονδίνο. Δεν μπορώ να απαντήσω απευθείας αυτή την ερώτηση, διότι αυτό πιστεύει η Coca-Cola. Γι' αυτό λάβατε αυτή την απόφαση να στερήσετε την Ελλάδα από 13 εκατομμύρια δολάρια σε αυτή την τόσο δυσχερή θέση στην οποία βρισκόταν. Κοιτάξτε, αυτό που κατανοώ εγώ είναι ότι πηγαίνοντας στην έδρα στην Ελβετία μπόρεσε η εταιρεία να έχει πρόσβαση στις χρηματαγορές και καλύτερη πρόσβαση. Γιατί οι χρηματαγορές στις Ηνωμένε Πολιτείες δεν έχουν την ίδια αξία το Zoom είναι που σας έκανε τη διαφορά. Έτσι είχατε καλύτερη πρόσβαση στις χρηματαγορέ, Αυτό θέλετε να πιστέψουμε. Πιστεύω ότι και οι ταξιογραφέ από τις αμερικανικές χρηματαγορέ μετακινήθηκαν. Έτσι κατάλαβα κι εγώ. Θέλατε, αυτό μας είπατε εσεί τουλάχιστον. Πήγατε στο Zoom για να έχετε καλύτερη πρόσβαση στι χρηματαγορέ, έτσι. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και τώρα η Walt Disney. Ευχαριστώ. Βλέποντας με τη σειρά τα ερωτήματα. Το πρώτο αφορούσε την πληρωμή των συμβούλων. Φυσικά θα σας δώσουμε αυτές τις πληροφορίες όπως το ζητήσατε. Οι τα περισσότερα κόστη μας για τη φορολογία αφορούν τη συμμόρφωση και το ότι έχουμε δραστηριότητες σε πολλές χώρες. Γι' αυτό δεν ξέρουμε απαραίτητο τα πάντα εκ των προτέρων για κάθε χώρα. Αλλά θα σας δώσουμε την πληροφορία. Τώρα για, τις, για τα δάνεια μεταξύ εταιριών. Δεν γνωρίζω να έχουμε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο εξάλλου και το CCCTB όπως και το BEPS, θα τις κλείσουν αυτές τις δυνατότητες. Και αυτό νομίζω ότι θα είναι καλό. Και τέλος, για την ετικέτα δίκαια φορολόγηση. Σωστό μου φαίνεται και αυτό. Αλλά όταν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρχουν αντικειμενικότατα κριτήρια και αν γίνει έτσι τότε νομίζω ότι θα ήταν για τους καταναλωτές και τις καταναλώτερες πολύ σημαντικό. Κυρία Γέιτς τώρα, του Μακδόναλντ. Για να προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις που αφορούσαν τον Μακδόναλτ η επιθετική λέει φοροαποφυγή. Η McDonald's πληρώνει ψηλούς επιχειρησιακούς φόρους και η ίδια η εταιρεία και όσες αδειοδοτούνται από μας. Ε, γύρω στα 32-33% στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη περίπου το 20, ε, κατά μέσο όρο 27% τα τελευταία 5 χρόνια. Τρία τέταρτα της δουλειάς μας στην Ευρώπη γίνεται με τις αδειοδοτήσεις βέβαια. Τώρα, για τον σχεδιασμό της φορολόγησης του McDonald's. Όχι, δεν βασιζόμαστε στο κέρδος, αλλά στη συμμόρφωση της επιχείρησης με τον, τους ισχύοντες νόμους. Αν γίνει αναδιάρθρωση, δεν έχουμε εμείς τις κυρίες ιδέες, απλώς μας συμβουλεύονται. Τώρα για το ποσά τις αμοιβέ που δίνουμε στους συμβούλους. Έχουμε μικρό προσωπικό σε ορισμένες αγορές και θα προσπαθήσω να τα συνδυάσω όλα αλλά πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς ζητάτε. Εμείς πληρώνουμε τους εξωτερικούς μας συμβούλους, τους ελεγκτές και ένα τμήμα του προπολογισμού μας είναι γι' αυτό. Αν μπορείτε να μας αποσαφηνίσετε το ερώτημα θα σας τα βρω. Θεωρούμε αυτές τις αμοιβέ πολύ σωστές. Δεν έχουμε το ίδιο σύστημα με την Coca-Cola για μερικές, μερικούς τομείς όπως τους φόρους για κτίρια χρησιμοποιούμε την ίδια μέθοδο στη ΣΥΠΑ αλλά όχι αλλού. Πού είναι τώρα γιατί το έχασα. Mm. Για το Λουξεμβούργο είχα πει ότι υπάρχουν μερικά προκαταρκτικά συμπεράσματα σε μια από τις εκθέσεις που ονοματίστηκε που έλεγε ότι ο κύκλος εργασιών και όχι το κέρδος έχει υπολογιστεί διαφορετικά. Πρέπει να ξέρουμε ότι τα, οι συμμετέχουν στη φορολόγηση γιατί υπάρχει το θέμα των δικαιωμάτων. Έχουμε εταιρείε που χρησιμοποιούν διεπιχειρησιακά δάνεια και τα επιτόκια που επιβάλλουμε είναι αυτά που ισχύουν στην αγορά. Τα υβριδικά εργαλεία δεν τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, μπορεί και καθόλου. Αλλά για τη σαφήνεια εμείς δίνουμε συμβουλές γιατί θέλουμε να συμμορφωθούμε με τον νόμο. Και το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε ισοτιμία, δίκαιος ανταγωνισμός είναι κάτι πολύ ουσιώδες για τις μεγάλες και μικρές εταιρείες και σε εμάς ε, υπάρχουν και τα δύο είδη. Η ετήσια μελέτη τώρα, επειδή πληρώνουμε τόσο πολλούς φόρους, δεν είμαι βέβαιη ότι γνωρίζω από πού προέρχεται αυτό, αλλά τα παίρνουμε όλα σοβαρά και πληρώνουμε όλους τους φόρους που χρωστάμε. η ετικέτα της δίκαιας φορολόγησης ακούγεται σαν πολύ σωστή ιδέα, αλλά ποιος θα αποφασίσει πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί. Γιατί το πόσο φόρο πληρώνεται εξαρτάται από το που λειτουργείται. Αν υπάρχει μία ένας ενιαίος φορολογικός συντελεστής στην Ευρώπη, μπορεί να είναι πιο εύκολο να αποφασιστεί αυτό. Αν όμως μπορούν οι χώρες να ανταγωνίζονται για τους συντελέστέ με διαφορετική βάση, τότε μπορεί να μην είναι τόσο σίγουρο αν μπορεί κανείς να καταλάβει α, κατά πόσον είναι δίκαιο. Σας ευχαριστώ. Εγώ. Τι λέει η Ινμπεύ. Έχει να προσθέσει τίποτα. Με ευχαριστώ. Να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Κάπελ για την ενιαία βάση φορολόγηση επιχειρήσεων και ε, την, ε, το transfer pricing, τη μεταφορά ε, τιμολόγησης. Αυτό θα απλουστεύσει τα πράγματα, θα μειώσει τους κινδύνους διπλής φορολόγησης. Και έτσι θα μπορούμε να έχουμε και ένα σύστημα πιο προβλέψιμο και πιο μόνιμο, ε, φορολογικό. Αν αναβληθεί αυτή η ενοποίηση της φορολογικής βάσης του CCTP, πράγμα που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει κίνδυνος να συνεχίσει η διπλή φορολόγηση κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος. Θα είναι τεράστιο πρόβλημα και παράληψη αυτό. Δεύτερον, εάν, συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος, αυτό τι σημαίνει. Ζητάτε μάλλον να περάσουμε ε, απευθείας στην ενοποιημένη φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις. Ακριβώς. Και το δεύτερο, για να επανέλθουμε στη συζήτηση που είχαμε για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα παγκόσμιο ανταγωνισμό εκτός των συνόρων. Εάν η κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ο φορολογικός συντελεστής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν βαθμό που θα είναι πολύ υψηλότερο από τον πραγματικό φορολογικό συνεργαστή σε αγορές ανταγωνιστικές για τις επενδύσεις, αυτό ενδεχομένω να έχει αρνητική επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα και καλό θα ήταν να το έχουμε και αυτό υπόψη μα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα θα δώσω το λόγο στους τελευταίους ε, βουλευτές. Ο κύριος Τόμ Φαντακάντελάρα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά χρειάστηκε αρκετό χρόνο για να σα φέρουμε στο κοινοβούλιο, αλλά χαίρομαι που σα βλέπω απόψε εδώ και πραγματικά είχε οριμάσει η κατάσταση για να μην πω τίποτα χειρότερο. Ε, το ακούσαμε σήμερα αυτό ε, ότι εταιρείε που είναι πολυεθνικές χωρίς καμιά σχεδόν εξαίρεση ψάχνουν να βρουν κατασκευάσματα ε, και τρόπους να πληρώνουν λιγότερους φόρους. Πρέπει ε, να έχετε ένα επιχειρηματικό μοντέλο, δεν διαφωνώ, αλλά πολλαπλασιάζονται ε, αυτά ε, τα συστήματα, τα κέρδη, δίνεται μερίσματα, θέλουν οι μέτοχοι περισσότερη απόδοση και εξαρτώνται από τους μετόχους οι εταιρείες σας για τη χρηματοδότηση. 55 δισεκατομμύρια ε, ε, βγήκε ένα ομολογιακό δάνειο για την ΙΜΠΕΒ όταν αγόρασε ε, μία άλλη εταιρεία και άρα όταν υπάρξει μια εναρμόνιση και κανόνες ίδιοι για το παιχνίδι δεν θα είναι έναν υπέρβλητο εμπόδιο για σας. Η μόνη λύση είναι το CCCTB ή πρέπει να λάβουμε και άλλα στοιχεία υπόψη μας. Εσείς τι λέτε. Και ποιος είναι ο συντελεστής που θεωρείται ε, δίκαιο για να το πληρώνετε. Και θα ήσασταν υπέρ μιας ενιαίας, ενός ενιαίου συντελεστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεωτικού για όλες τις εταιρείες. Και ναι, και πάλι ποιο θα ήταν το ύψος αυτό το ιδεώδης για σας. Όλε Λούτβιξον, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ. Έχω μια-δυο ερωτήσει για τον κύριο Μάτσον. Της IKEA. Δεν αναφέρομαι μόνο στην IKEA, αλλά στις εταιρείε όλου του ομίλου. Ως προς τους φόρους, ξέρουμε ότι είσαστε μια από τις εταιρείε με τον επιθετικότερο φορολογικό σχεδιασμό παγκοσμίω. Έχω λοιπόν μια ερώτηση για το LuxLeaks που εκτεθήκατε κι εσείς. Έχετε ένα ίδρυμα με έδρα στο Λιχτενστάιν και την Ολλανδία και την εταιρεία Holding στο Λουξεμβούργο, την IKEA Holding SA. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της εταιρείας Holding πέρα από το να έχετε τον χαμηλότερο δυνατό φόρο. Εάν δεν έχετε μια πολύ γενναιόδορη συμφωνία με τον Λουξεμβούργο και τις αρχές του, θα είχατε διαλέξει αυτό το είδος την ε, διθέτηση, τη διοργάνωση. Και η δεύτερη οργάνωση έχει να κάνει με τις πρόσφατες εξελίξεις γενικότερα. Με το LuxLeaks, με το γεγονός ότι θα μειωθεί η κρατική βοήθεια, ότι οι καταναλωτέ διαμαρτύρονται κατά των ε, φορολογικών συμφωνιών έχουν ληφθεί κάποια πολιτικά μέτρα ε, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τι συμπέρασμα αντλείται από αυτές τις εξελίξεις. Υπάρχει περίπτωση ο φορολογικός σας σχεδιασμός να γίνει λιγότερο επιθετικός. Έχετε εξηγήσει ότι δεν σας νοιάζει. Έχετε δηλώσει ότι δεν σας νοιάζει πως αντιδρά ο κόσμος. Δεν θα αλλάξετε τίποτα. Είναι σωστό αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Νίδα Μαγιά, ξαναρχόμαστε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ. Δύο μάλλον τεχνικές ερωτήσεις. Ε, και κάπω πολιτικές. Οι εταιρείε σας, αναρωτιέμαι. Αν η συζήτηση γινόταν για το CCTV, θα μπορούσαν να μας πούνε ξεκάθαρα ότι είναι υπέρ. Είστε Είπε, ή προτιμάτε να έχετε και κάποια εναλλακτική λύση. Δεύτερον, συμφωνείτε όλοι με το συνάδελφό σας που είναι υπέρ του CCCTB και όχι CCTB, δηλαδή είναι ενοποιημένη βάση, όχι απλώς κοινή. Και για το CBCR, που είναι η αναφορά αναχώρα ε, στους ισολογισμούς, τι πληρώνεται κάθε φορά. Ξέρετε ότι αυτή η συζήτηση κυριαρχεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι μόνο λοιπόν η αναφορά αναχώρα, ε, ε, αν θα πρέπει να γίνεται ή αν θα πρέπει να είναι δημόσια η υπόθεση αυτή, να τα γνωρίζουν μόνο οι εφορίες. Γιατί αν είναι εντελώ δημόσια αυτά για το γενικό κοινό, υποχρεώνονται κάποιε εταιρείε ε, να αποκαλύπτουν κάποια στοιχεία που δεν αποκαλύπτουν οι ανταγωνιστές. Ε, τι λέτε λοιπόν για τη φορολογική σας ε, δήλωση αναφορά κατά χώρα. Είναι στοιχεία ευαίσθητα και πρέπει να είναι αυτά εμπιστευτικά ή όχι. Τελευταίο ο Πέτερ Ζήμων από σοσιαλιστέ και δημοκράτε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση προς όλους καταρχάς, προς όλες τις εταιρείες που έχουμε εδώ ενώπιόν μας. Είμαι βέβαιος ότι θα έχετε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει δημοσιεύσει ένα κατάλογο τέλη Ιουνίου για τους φορολογικούς παραδείσους. Οι εταιρείε σας έχουν ελέγξει αν σε αυτές τις χώρες που αναγράφονται εδώ έχετε θηγατρικές και παραρτήματα. Εάν ναι, σας ερωτώ ποια είναι αυτά και ποιες δραστηριότητες ασκείτε εκεί σε τι βαθμό και πόσο προσωπικό εργάζεται εκεί. Άλλη ερώτηση. Για τον Για την... Ε, ε, το 2014, 1,5 δις κέρδη δηλώσατε InBev και πληρώσατε μόλις 1% φόρους. Και αυτό ε, μπορεί να αναχθεί ε, στο ruling ε, του υπερβολικού κέρδους. Αυτό αφήνει αφορολόγητες κάποιες ενδομήλικες συναλλαγές. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε πώς φτάσατε σε αυτή τη μείωση. Γιατί εγώ δεν ξέρω καμία εταιρεία στον πραγματικό κόσμο που να έχει τέτοια φοροαπαλλαγή και να έχει τόσα κέρδη που να έχουν προκύψει από συνέργειες μεταξύ των εταιριών. Και αν δεν είναι το 99% να είναι και 60% και 50% και 40%. Να μου το εξηγήσετε στη βράξη για να δω πώς... Δεν ξέρω καμία εταιρεία που να λειτουργεί έτσι. Μου φαίνεται τελείως ακατανόητα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο τώρα ε, με την αντίστροφη σειρά στους προσκεκλημένους. Να αρχίσουμε από την ΙΝΠΕΒΑ και Νόιζερ Μπούς. Τις δηλαδή. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα απαντήσω με τη σειρά. Στην ερώτηση του κυρίου Βαντεκέντελαρ, Θα ήθελα να πω πως η σημασία προσδίδουμε στη Σύμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διατησία για να υπάρξει ένας πιο εύκολος τρόπος και πιο απλός για την επίλυση των διαφορών. Αυτό είναι για μας προτεραιότητα. Και θέλουμε ιδιαίτερα να εστιάσουμε σε αυτή. Γι' αυτό που ρώτησε ο κύριος για ε, την ενιαία φορολογική βάση ή φορολογική βάση. Για μας είναι πολύ σημαντικό να είναι ενοποιημένη αυτή η φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις, να είναι CCCTB και όχι απλώς CCTV και για την αναφορά αναχώρα. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Και βεβαίως θα το καλωσορίζουμε αυτό, να αναφέρονται οι φόροι αναχώρα. Είναι σημαντικό εργαλείο αυτό για τις φορολογικές αρχές για να καταλαβαίνουν καλύτερα πώς λειτουργούν φορολογικά οι πολυεθνικές εταιρείες. Είμαστε κατά όμως της δημοσίευσης ε, της ε, πληροφορίας αυτής χώρα. Εγώ μιλώ μόνο για τη δική μας εταιρεία και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούμεθα και δεν μπορώ να μιλήσω εξ άλλων, αλλά ανησυχούμε γιατί αν μας ζητήσουν τέτοιες πληροφορίες και αυτές μπορούν να συνδυαστούν με άλλες δημόσιες, αυτό μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητο και να αφορά εμπορικά απόρριτα σε σχέση με ανταγωνιστές μας. Ανισχούμε πάρα πολύ λοιπόν. Ε, σε περίπτωση που δημοσιευθούν αυτά τα στοιχεία υπάρχει κίνδυνος και υπονομεύει αυτό την ανταγωνιστικότητα σίγουρα στο δικό μας κλάδο. και ο τρόπος με τον οποίο να ανταλλάσσουν πληροφορίε, οι εφορίες και οι διάφορες φορολογικέ αρχές θα πρέπει να είναι πάρα πολύ εξασφαλισμένος με ε, δικλείδε έτσι ώστε να μην διαραίουν αυτά τα στοιχεία να μην δημοσιεύονται. Ε, για την ερώτηση τη ερωτήσεις του κυρίου Ζήμων ε, για, για τους φορολογικούς παραδείσους. Είναι απλούστατη η απάντηση. Εμεί δεν είμαστε παρόντες σε φορολογικού παραδείσους για φορολογικού ε, λόγους. Αφήστε δε που ε, ελέγχεται και ο ορισμός ε, του φορολογικού παραδείσου. Μα υπάρχει λίστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέει ο κύριο Ζήμων. Εντάξει, αυτά λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά άλλοι έχουν άλλες λίστε ε, θα πρέπει κάπως να οριστεί διεθνώς η έννοια του φορολογικού παραδείσου. Για μας λοιπόν είναι σαφής η πολιτική, εμείς πληρώνουμε τους φόρους μας εκεί που παράγουμε κέρδη και βεβαίως έχουμε σε κάποιες χώρες ε, εταιρείε που μπορεί να θεωρούνται φορολογική παράδειση χώρες για διάφορους λόγους και ιστορικούς, γιατί αγοράσαμε εταιρείε που είχαν ε, ε, κάποια εργοστάσια πολλές φορές μπορεί πλέον να μην χρειάζονται ή να μην χρειάζονται για φορολογικούς λόγους, αλλά δεν είναι εύκολο να φύγεις πάντα από μια χώρα. <laughs> Και καμιά φορά είναι πολλά τα νομικά εμπόδια και τα διοικητικά για να σηκωθεί να φύγει τελείω από ένα φορολογικό παράδεισο. <laughs> Um, και ξέρετε, παρόντες είμαστε παντού και όχι για φορολογικού λόγους και σε φορολογικού παραδείσους μπορεί να είμαστε γιατί πουλάμε μπύρα και πίνει ο κόσμος μπύρα. Αλλά το πρώτο, μα τι κάνετε ε, για να πληρώνετε τόσο λίγους φόρους. Το θέμα δεν είναι ότι πίνουν μπύρα οι ανθρωπικοί και τους αρέσει η μπύρα σας, αλλά για λόγους οικονομικούς έχετε πάει. Αν δεν είμαστε παρόντες, και παραμένουμε για λόγους ιστορικούς, γιατί αγοράσαμε ρε παιδί μου μια εταιρεία κάποτε που ήταν παρούσα εκεί και είχε μια φορολογική κατασκευή, αλλά πλέον αυτό έχει εγκαταληφθεί. Και είναι στα βιβλία τα φορολογικά και δεν, δεν έχει καμία δραστηριότητα. Το είπαν και άλλοι, για να το απλοποιήσουμε, προσπαθούμε να μειώσουμε τις εταιρείε που συμμετέχουν στον όμιλο, αλλά δεν είναι πάντα απλό και εύκολο αυτό. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πάντα και τις πρακτικές και τις πραγματικές ε, συγκυρίες. να μιλήσω για το βελγικό ζήτημα, δεν έχω χρόνο. Το 1% βασίζεται σε μια βασική παρανόηση, παρεξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο φορολογείται η εταιρεία μας. AB InBev SA. Είναι η βελγική εταιρεία και τα κέρδη προέρχονται από μερίσματα από τους ομίλους και αυτά στο Βέλιο είναι αφορολόγητα τα μερίσματα έχουν φόρο απαλλαγή εξού και το 1% φόρο που πληρώνουμε Je vous remercie. Ευχαριστώ κυρία Μακδόναλτ. Ως ό,τι αφορά τους ισότιμους κανόνες, ναι, νομίζω ότι είναι απαραίτητη. Η ερώτηση αφορούσε το τι γίνεται στην Ευρώπη, αλλά εμείς είμαστε μια διεθνής πολυεθνική. Έχουμε και την αμερικανική πολιτική και τις φορολογικές απαιτήσει εκεί. Εφόσον μπορούσαν όλα να εναρμονιστούν, αυτό θα ήταν λίγο φιλόδοξο. Μένει πολύ καλό, θα μας βόλευε. Ε, πολύ θα ήθελα και οι McDonald's και οι franchisers να λειτουργούν σε όλες τις χώρες και να πληρώνουν σωστά τους φόρους, αλλά είναι εταιρική ευθύνη οι φόροι και εφόσον τα ποσά που συγκεντρώνονται δαπανώνται σωστά, δεν μπορούμε να προτείνουμε εμεί ενίο συντελεστή. Από την άλλη, έχουμε πολλές ανησυχίες για την ε, διατησία της, την επίλυση διαφορών. Ήδη υπάρχουν κάποιες υποθέσεις, ε, κάποιες φορέ μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, με άλλες χώρες, αλλά οτιδήποτε μπορεί να βελτιώσει την φορολογική σταθερότητα θα εκτιμηθεί. Για τις σχετικές βοήθειες του LuxLeaks και τις σχετικές αποκαλύψεις, η McDonald's έχει 8.000 εστιατόρια στην Ευρώπη δεν αλλάξαμε ή μετατρέψαμε την δραστηριοποίησή μας εξαιτίας αυτού του σκανδάλου. Πιστεύουμε ότι πληρώνουμε σωστά τους φόρους, είναι και σημαντικά τα ποσά και το κάνουμε και με μεγάλη μας χαρά. Είμαστε υπέρ του CCCTB, αλλά για να επαναλάβω κάτι που είπαν και οι υπόλοιποι υποστηκλημένοι, θα πρέπει αυτό να είναι και συνεπές και σαφές το σύστημα. Για την υποβολή εκθέσεων αναχώρα, κανένα πρόβλημα, αλλά για την αποκάλυψη των πληροφοριών της εταιρεία δημοσίω μας ανησυχεί και το φοβόμαστε. Να μοιραστούμε τις πληροφορίες μας με τις εφορίες όταν μας ζητούνται με κάποιο αίτημα συγκεκριμένο, ευχαρίστως θα συνεχίσω να το κάνω, αλλά ο κίνδυνος παραπληροφόρησης, ο κίνδυνος σύγχυσης περίπλοκων λεπτομεριών, και ε, πληροφορίες που μπορεί να είναι ευαίσθητες για την ε, ύπαρξη της εταιρεία είναι πολύ δύσκολο. Άλλο να τις παίρνουν φοροτεχνικοί και εφορίες, αυτοί που τα καταλαβαίνουν κάπως διαφορετικά και τους αφορά στη δουλειά τους, ναι, αλλά άλλο το κοινό. για τον κατάλογο φορολογικών παραδείσων της Ευρωπαϊκής Ένωση. Όπως πίνουν μπύρα οι άνθρωποι, ελπίζουμε ότι και χάμπουργκερ θα συνεχίσουν να τρώνε και τα άλλα προϊόντα της McDonald's. Έχουμε κάποιε εταιρείε σε χώρε φορολογικού παραδείσου, αλλά οι επιχειρηματικέ μα δραστηριότητε εκεί έχουν να κάνουν και με τα εστιατόρια και τη λειτουργία του και κάποιε περιπτώσει management αποκεντρωμένου. Τα καταστήματα, τα εστιατόρια ε, in franchises είναι τοπικό, σε, οργανωμένοι σε τοπικό επίπεδο. Έτσι λειτουργούν και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Σα ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Στόουαλ. Ευχαριστώ. Πολλά τα ερωτήματα. Ελπίζω να μπορέσω να τα απαντήσω όλα. Το πρώτο αφορούσε τα BEPS. Ξέρω και καταλαβαίνω τις ανησυχίες για τις τεχνη, τους τεχνητούς φορολογικούς διακανονισμούς. Αλλά εμείς δεν κάνουμε τέτοια κόλπα. Παραδείγματο χάρη όταν ε, στέλνουμε πληρωμές στη ΣΥΠΑ για μας είναι αντικίνητρο. Ζητάμε δηλαδή μια μείωση σε άλλες χώρες σε ρυθμό χαμηλότερο από αυτόν τον οποίο πρέπει να πληρώσουμε μετά στη ΣΥΠΑ. Και η φορολογία στην Αμερική τα προσέχει πολύ αυτά. για το CCCTB. Νομίζω ότι θέλουμε πρώτα να δούμε τις λεπτομέρειες, να δούμε πώς ακριβώς θα υπολογίζεται για να μπορέσουμε να απαντήσουμε ειλικρινά. Και ορισμένες από τις σκέψεις που ανέφερε και η Coca-Cola είναι από εκείνες που πρέπει πρώτα να αναλύσουμε πριν να πούμε αν είμαστε υπέρ ή κατά. Αλλά αν όμως γίνει δίκαια και πρακτικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην οικονομία της επιχείρησης και κατανέμονται σωστά τα κέρδη της επιχείρησης μεταξύ χωρών, τότε για μας θα ήταν θετικό γιατί θα απλοποιούνταν η διαχείριση της φορολογίας. Τώρα κατά πόσο χρειάζεται ενιαίο συντελεστής. Δεν είμαι εμπειρογνώμων αλλά θα έλεγα ότι Ο συντελεστής προφανώς δημιουργεί φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ κυβερνήσεων οι οποίες προσφέρουν κίνητρα για διάφορους λόγους για να προσελκύσουν οικονομική δραστηριότητα. Είναι λοιπόν κάτι που θα επηρέαζε τη συμπεριφορά της επιχείρησης, αλλά θα το αφήσω αυτό στους ειδικού. Για τις εκθέσεις χώρα με χώρα, και κατά πόσο πρέπει να είναι δημόσιες αυτές οι πληροφορίες, συμμερίζομαι τις ανησυχίες και μερικών άλλων εταιριών. Τα μέλη του ΩΣΑ βασικά κατέληξαν σε μια πολύπλοκη συμφωνία για αυτό το εργαλείο αξιολόγησης υψηλού κινδύνου μεταξύ φορολογικών αρχών οι οποίες αποκαλύπτουν μεγάλο ποσοστό των πληροφοριών τους και των δραστηριοτήτων τους μέσω των επισήμων εκθέσεών τους. Και υπάρχει μια πολύ λεπτομερέστερη ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ φορολογικών αρχών των χωρών όπου λειτουργούμε και εμπειρογνώμονες τα εξετάζουν όλα αυτά για να είμαστε βέβαιοι ότι συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους στην κάθε χώρα. Κατανοώ τις ανησυχίες για τα περιθώρια αποκαλύψεων και λοιπά και κατά πόσο θα έπρεπε αυτά να είναι δημόσια έγγραφα ή όχι. Αν όμως το απαιτήσουν οι κυβερνήσεις, φυσικά θα συμμορφωθόμεν. Τώρα για το τελικό ερώτημα που έχω εδώ για τους φορολογικούς παραδείσους και σε άλλες ακροάσεις εδώ μέσα δεν βρέθηκε κοινό ορισμός περί του τι είναι φορολογικός παράδεισος. Καμιά φορά ας πούμε το Hong Kong άδικα κατ' θεωρείται φορολογικός παράδεισος αν και έχει πολύ μεγάλη οικονομική δραστηριότητα και πληθυσμό. Και εμείς έχουμε δραστηριότητες στο Hong Mong. Και ξέρουμε ότι παίζουμε σε κάποιο σημαντικό ρόλο και Και φυσικά ε, και στις Μπαχάμες έχουμε αναγκαστεί να ιδρύσουμε μια τοπική εταιρεία για να μπορούμε να δράσουμε εκεί. Σε μερικές χώρες απαιτείται αυτό το πράγμα για προφανείς λόγους, αλλά το κυριότερο που πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι τα κέρδη μας αφήνουν πάντα κάποιο οικονομικό ίχνος και ας πούμε ότι κάποια εταιρεία αγοράζει κάποια άλλη που βρίσκεται σε κάποιο λεγόμενο φορολογικό παράδεισο αλλά με πολύ λίγη δραστηριότητα. Εδώ το θέμα θα ήταν δημιουργούνται εκεί σημαντικά κέρδη ή όχι. Και δεν υπάρχει επομένως και λόγος σημαντικής φορολόγησης. Αν έχετε μία υπνότουσα οντότητα στα νήσους Καϊμάν, φυσικά δεν θα φορολογηθείτε και πολύ Βέβαια το να μην έχει δραστηριότητα αλλά να εμφανίζει σημαντικά κέρδη θα ήταν πρόβλημα λοιπόν. Εμείς ξέρουμε πάντως και είναι γνωστό πού πληρώνουμε φόρους και συνδυάζονται σαφώς με τις αληθινές οικονομικές μας δραστηριότητες. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Coca-Cola. Bob Jordan. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman, <clears throat> thank you for the questions. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ένα σχόλιο επαναλήφθηκε μεταξύ των ερωτήσεων για το CCTB και η ερώτηση ήταν αν είναι αυτός ο μόνος τρόπος για να υπάρξουν ισότιμοι κανόνες. Και εάν χρειαζόμαστε έναν και μόνο φορολογικό συντελεστή. Μια άλλη ερώτηση ήταν αν θα προτιμούσαμε το CCTB να χρησιμοποιηθεί αντί για το CTV και αν θα θέλαμε να είναι δημόσιο ή μη το ποσοστό αυτό. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπο να δημιουργηθούν ισότιμοι κανόνε. Ε, νομίζω ότι θα μπορούσε μάλιστα να συμβάλλει σε αυτόν τον σκοπό βέβαια, αλλά είναι πιο περίπλοκο το θέμα. Είναι δύσκολο να είναι εναρμονισμένη η βάση και να ισχύουν οι σωστοί παράγοντες. Θα είναι πολύ δύσκολο ακόμη και να ορίσουμε τον όμιλο στο σύνολό του. Αλλά ακόμη και μέσα στον ίδιο τον όμιλο κάποιες εταιρείε διευθύνονται από διαφορετικά τμήματα του ομίλου με μεγαλύτερο, μεγαλύτερο περιθώριο από ό,τι άλλες. Και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πέραν των άλλων διαφορών μεταξύ των διάφορων τμήματων δραστηριοποίησής μας. Πάντως, με την πρωτοβουλία BEPS και με όσα έχει κάνει και η Επιτροπή σας, θα μπορούσαμε να οδεύσουμε προς ένα σύστημα ισότιμων κανόνων. Η με της το πρόγραμμα δράσης στα σημεία ενός 10 η υποβολή εκθέσεων αναχώρα, όλα αυτά θα μπορούσαν να ενισχύσουν το, το σύστημα με τους ισότιμους κανόνες, αλλά <clears throat> είναι και η επίλυση διαφορών κάτι το σημαντικό. Θα βοηθούσε, διότι ασχέτως του πόσο απλούς νόμους προσπαθούμε να σχεδιάσουμε, πάντοτε θα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που περιπλέκουν την κατάσταση. Η ρήτρα για την επίλυση διαφορών με την υποχρεωτική διατησία ίσως να μην σημαίνει ότι οι διαφορές πάνε κατευθείαν στο διατητή για επίλυση. Απλώς ότι ε, η διαφορά μπορεί να επιληθεί σε μια από τις προγενέστερες φάσεις της διαδικασία, εφόσον το θέλουν ε, τα δύο μέρη απλώς ο διατητής θα ε, είναι η λύση όταν χρειάζεται περισσότερη συζήτηση μεταξύ των δύο για το CCTB και αν το χρησιμοποιούμε έναντι του CCTB υπάρχουν πολλές επιπλοκές εδώ ε, και πολλές δυσκολίες σε σχέση με το CCCTB. Ε, νομίζω θα επέλυε πιο πολλά θέματα από ότι το CCTB που διατηρεί πολλές από τις σημερινές δυσκολίες όπως την ε, μεταφρατμολόγηση το transfer pricing. Εάν έχει κανείς κοινή βάση, αλλά υπάρχει πάλι αυτό το θέμα της μεταβάσης τιμολόγησης, δεν αλλάζει κάτι. Για τον ε, κοινό φορολογικό συντελεστή, δεν μπορώ να το πω εγώ, αυτό θα το αποφασίσω, αλλά ξέρω ότι στην έκθεση της Επιτροπής σας λέγεται ότι ο φορολογικός σχεδιασμός πρέπει να γίνεται εντός των πλαισίων του νόμου και των ισχυουσών συνθήκων. Οπότε η καταλληλότερη απάντηση για τον ε, φορολογικό συντελεστή είναι η διεθνή συντονισμό και οι συνθήκε που ισχύουν και ε, θα πρέπει να υπάρξουν διαπραγματεύσει για να υπάρξει ένα συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο θα πρέπει να κατευθύνουν προ τη σωστή ε, κατεύθυνση τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουν εφόσον αυτό είναι ο σκοπό σα. Και τέθηκε και ένα θέμα για του καταναλωτέ που αρχίζουν να τα προσέχουν. Αυτά βεβαίω και ισχύει. Οι καταναλωτέ έχουν επιλογή ποιο αναψυκτικό θα επιλέξουν. Νομίζω ότι δική μας ευθύνη είναι να αποδεικνύουμε την αξία μας καθημερινά σε κάθε μια από τις τοπικές περιοχές όπου λειτουργούμε. Και για τους ε, φορολογικούς ε, κανόνες και το φορολογικό σχεδιασμό σε όλα τα κράτη-μέλη και σε πάνω από 200 χώρες που πουλούνται τα αναψυκτικά μας είναι πολύ σημαντικό την κοινωνική αποδοχή αυτή να τη διατηρήσουμε. Τώρα για τους φορολογικούς παραδείσους, τέθηκε και γι' αυτό ένα ερώτημα. Η φορολογική παράδειση ορίζονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Πάντως, γενικώ φορολογική παράδειση έχουν χαμηλό φορολογικό συντελεστή και όπως είπα προηγουμένως και σε εσά πρόεδρε με την ερώτησή σας για τον πρόσθετο φόρο που θα έπρεπε να καταβάλουμε ως αμερικανική εταιρεία όταν τα περισσότερα κατευθύνονται πάλι προ τι ΗΠΑ χρησιμοποιούμε τι εταιρείε holding ώστε να μπορούμε να επανεπενδύσουμε τα κέρδη από τις ε, δραστηριότητες μας εκτός Αμερικής στις ε, χώρες όπου λειτουργούμε, στις συγκεκριμένες κοινότητες. Οπότε έτσι εξυπηρετείται και ένας σκοπός. Και όπως ε, ο συνάδελφος την InBev και την McDonald's και την Disney έχουμε καταναλωτές σε πολλές χώρες, χώρες που θεωρούνται φορολογική παράδοση, αλλά και δραστηριοποιούμαστε εκεί και πολλούς απασχολούμε και πολλά κεφάλαια επενδύουμε στις χώρες αυτές που μπορεί κατά τα άλλα να θεωρούνται και φορολογική παράδειση. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάτσον. Ευχαριστώ. Έχω πολλά προφανώς να πω γιατί τέθηκαν πολλά ερωτήματα αλλά για την υποβολή εκτός είναι ένα χώρα. είμαστε υπέρ. Έχουμε τοπικές πληροφορίες, έχουμε τις ετήσιες εκθέσεις μας, πάρα πολλές λεπτομέρειες. Χρειάζεται βεβαίως καλύτερη διοργάνωση να ε, ενισχυθεί το σύστημα για να μπορούμε να υποβάλουμε τις σχετικές πληροφορίες στις ενδιαφερόμενες εφορίες. Αλλά μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το φόρτο. Θα έχουμε 160 παραπάνω εκθέσεις, οπότε να θυμίσουμε και στις εφορίες ότι πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα να τα καλύψουν αυτά. Διότι Βεβαίω θα αυξηθεί και η δική του δουλειά και ο δικό του φόρτο εργασία. Όμω πρέπει να υπάρχει αυτή η υποβολή εκθέσεων χώρα. Τώρα, για την ενοποίηση τη φορολογική βάσης είμαστε βεβαίω υπέρ, αλλά θα έπρεπε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση παρέκκληση, δηλαδή να συμφωνήσουν όλοι. Να μην δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει ή διαφορέ μεταξύ των χωρών. να μην χρειάζεται να πάμε στις φορολογικές αρχές απαραίτητο. Μιλώντας τώρα για τον ΟΣΑ και το transfer pricing και τις κατευθύνες γραμμές του ΟΣΑ, βεβαίως μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα και για μας. Όμως η κοινή βάση είναι κάτι που το θέλουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μοιηθεί το διοικητικό άχθος, ε, αυτό είναι κάτι που θα μας εξυπηρετούσε. Επίσης για την ενοποίηση της φορολογικής βάσης. σε γενικές γραμμές δεν έχουμε πρόβλημα να το στηρίξουμε, αλλά πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό. Βλέπω και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν όμως, διότι το τι γίνεται με το φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των εφορίων των διάφορων χωρών. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην εκθέσουμε την εταιρεία στην, ε, ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών φορολογικών αρχών. Είναι πολλή δουλειά που πρέπει να κάνουμε για να παραμείνουμε σωστοί επιχειρηματίες εδώ. Θα μπορούσε βεβαίω να το σκεφτεί κανείς μακροπρόθεσμα. Κύριε Λούντφιξον. Η IKEA δεν είναι όνομα εταιρεία, είναι όνομα μάρκας, είναι σήμα. Υπάρχουν 12 άλλες εταιρείε στον Όμιλο ε, με τόσους εργαζόμενους, τόσα προϊόντα, τόσες ε, συναλλαγές. Δεν έχω πληροφορίες για όλες. Ε, Μπορεί να τα βρείτε στο ίντερνετ. Όμως για τους για την franchise βρίσκεται στην Ολλανδία και ανήκει στην Ιντερικαία. Αλλά δεν μπορώ να απαντήσω για άλλες εταιρείες. Απλώς δεν έχουμε ούτε επιδοτήσεις στο Λουξεμβούργο ούτε στο Λιχτενστάιν. Και διαβεβαίω γι' αυτό δεν έχει τέτοιο πράγμα εκεί. Περί... Πληρώνουμε περίπου 20% φόρο επί του εισοδήματος. Είμαστε την ίδια χώρα, κύριε Λούτριξον. Εάν όλο μα το εισόδημα πήγαινε στη Σουηδία, θα πρέπει να πληρώνουμε 22% φόρο. Κοντά σε αυτό είμαστε, αν τα πράγματα που σα έδωσα. Και για τους φορολογικούς παραδείσους. Δεν πηγαίνουμε σε εξωτικά νησιά. Έχουμε ε, τοπική διοργάνωση, όχι διασυνοριακή. Εκεί που έχουμε τα καταστήματά μας και εκεί που λειτουργούν οι, τα εργοστάσια μας. Τέλος, Τέλος να πω ότι έχουμε πολύ λίγε φορολογικέ συμφωνίε για να παραγραφώ σε αυτά που έλεγε ο κ. Λούτβιξον και αυτό που χρειαζόμαστε είναι σαφήνεια, σαφήνεια και τίποτε άλλο. Είναι πολύ περίπλοκο το σύστημα και γι' αυτό πραγματικά στηρίζω όσα κάνετε. Έχουμε προσπαθήσει τόσο πολύ να καταλάβουμε όλες αυτέ τι απαιτήσει που υπάρχουν από εμά. οπότε αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε αποτελεσματικοί και ανταγωνιστικοί. Είναι πολύ σκληρά τα πράγματα στην αγορά. Στηρίξτε μας. Σας παρακαλούμε, στηρίξτε μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σούστερ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρώτη ερώτηση ήταν αν το CCTV είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσουμε ίσους κανόνες παιχνιδιού. Δεν νομίζω. Το σημαντικότερο είναι να έχουμε σαφείς κανόνες ευσύνοπτους, να τους καταλαβαίνουν όλοι, όχι μόνο οι φορολογούμενοι αλλά και οι εφορίε, γιατί καμιά φορά δεν καταλαβαίνουν ούτε οι εφορίες τους ίδιους τους κανόνες. Mm. Θα πρέπει λοιπόν να λειτουργούν όλα αυτά αμφίδρομα. Ήδη είπαμε ότι για το CCCTB για να λειτουργήσει χρειάζεται ενιαίο φορολογικό συντελεστή και έχω φιλοσοφικό πρόβλημα αν συνδυαστεί με ένα patent box γιατί ε, αυτό κάπως αποδυναμώνει τον ε, κοινό ενοποιημένο συντελεστή φορολογική βάση μάλλον για ε, την φορολόγηση των εταιριών. Καλά, αυτά είναι προσωπικές μου φιλοσοφικές απόψεις τώρα για τον ενιαίο συντελεστή ε, είμαι υπέρ, όπως είπα και προηγουμένως, ενιαίου φορολογικού συντελεστού. Ε, κάποιοι, οι συνάδελφοί μου δεν αναφέρθηκαν σε ποσοστό. Αν θέλει η Ευρώπη να κάνει ενιαίο συντελεστή θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικός. Θα πρέπει να κοιτάξετε τις χώρες γύρω σας. <laughs> Εγώ θα έλεγα γύρω στο 20% αλλά δεν είναι δική μου η απόφαση, θα πρέπει να τα αποφασίσουν οι Υπουργοί Οικονομικών. Ε, ίσως ε, αν αυξηθεί ο ΦΠΑ είναι πολύ δύσκολο να προβληθεί αυτό και να γίνει δεκτό και να πουληθεί εντός εισαγωγικών. Αυτά για το συντελεστή. Τώρα, για την έκθεση αναχώρα και αν θα πρέπει να δημοσιεύονται τα στοιχεία ή όχι. Εμείς, όπως το είπα και στην εισαγωγή μου, θα ήμασταν υπέρ μιας διαφάνειας ανάμεσα στους φορολογουμένους και στις εφορίες. Τώρα υπάρχουν στοιχεία εμπορικού απορρίτου, δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτά έτσι και να τα ξέρουν και οι ανταγωνιστές. Τα περιθώρια κερδών είναι πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία ε, για το δικό μας κλάδο και μπορεί κανείς από κάποιες προφορίες να συνάγει κάποια συμπεράσματα που δεν θέλουμε να είναι δημόσια. Γιατί μπορεί αυτό να οδηγήσει και σε παρερμηνίες και δεν θα το θέλαμε κάτι τέτοιο. Και η τελευταία ερώτηση είχε να κάνει με το αν έχουμε εταιρείε σε φορολογικού παραδείσους κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς καμία. <laughs> Και ξέχασα μια ερώτηση για το τι λέει η κοινή γνώμη για τη φοροαπαφυγή και φοροδιαφυγή. Όλες οι εταιρείε ε, ενδιαφέρονται για την κοινή γνώμη και η δικιά μας δεν διαφέρει σε αυτό. Αλλά η Philip Morris International δεν έχει τέτοια πράγματα φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Θα σε ευχαριστούμε και τους έξι που δεχτήκατε να κάνετε αυτή την ανταλλαγή απόψεων μαζί μας Απαντήθηκαν σχεδόν όλα τα ερωτήματα και όσες δεν απαντήθηκαν προφορικά υποσχεθήκατε να μας απαντήσετε γραπτός. Σας ευχαριστώ όμως μέχρι το τέλος της εβδομάδας αν το κάνετε. Τώρα οι συγκητές μήπως θέλουν να καταλήξουν. Η Ελίζα Φερέρα πρώτη. Ναι. Θα μιλήσω στα πορτογαλικά. Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σημαντικά όλα αυτά που είπαμε και η ανταπόκριση των εταιριών στην πρόσκλησή μας εδώ για δημόσια ανταλλαγή απόψεων. Δημόσια. Θα είχα... Να θέσω και ένα τελευταίο ερώτημα για να το σκεφτούμε. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις IKEA, Facebook, Walt Disney, Google, Coca-Cola κάνουν τεράστια προσπάθεια διαφήμισης και marketing στη σημερινή πραγματικότητα όπου οι καταναλωτές πληρώνουν τα σπασμένα με του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού δεν θα ήταν καλύτερο να έχετε μια πολιτική διαφήμιση που να προβάλλει ότι πληρώνετε σωστά τους φόρους σας και αυτό να, προ... να χρησιμοποιείτε ως μέθοδο marketing. Θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά των πολιτών να ξέρουν ότι οι μεγάλες πολυεθνικές πληρώνουν σωστά τους φόρους και όσα δαπάνες προσπαθούμε με τους εθνικούς προπολογισμού και τον ευρωπαϊκό προπολογισμό καλύψουμε. Αντί λοιπόν να χαλάτε χρήματα σε διαφημίσει τυχαία, να κάνετε μια διαφήμιση για τη διαφάνεια του ομίλου, για την εντιμότητα την εταιρική που να απευθύνεται στους πολίτες. Οι διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα αυτή της ακρόασης είναι συμπεράσματα που θα τα διεξαγάγουμε αργότερα. Απλώς νομίζω ότι μπορούμε να αποφανθούμε ότι υπάρχει ε, ουσιαστική διαφορά Ε, μάλλον υπάρχει ένα ε, ουσιαστικό σημείο στο όσο είπαν όλοι, ότι όλοι πληρώνουν τους φόρους εκεί που δραστηριοποιούνται. Κάτι που είναι σημαντικό με τις αδύναμες φορολογικές διαθετήσεις που υπάρχουν σε φορολογικούς παραδείσους ε, και τελικώς δεν είχαμε και επαρκείς εξηγήσει για αυτές τις περιπτώσεις. Εάν σας τα κατάλαβα και το επιχείρημα για τους υψηλούς ε, φόρους των ΗΠΑ, έτσι δημιουργείται μια κατάσταση που βεβαιώνει και το δική μας προηγούμενη διαπίστωση ότι πράγματι ε, κάποιες, κάποια εισοδήματα που θα έπρεπε να φορολογούνται ουσιαστικά παρκάρονται εντός ε, εισαγωγικών στις νήσους Κάιμαν, στις Βερμούδες, αλλού όπου δεν καταβάλλονται φόροι, πουθενά, σε καμία περίπτωση, οπότε αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα ως προς την ισορροπημένη κατανομή του φρολικού βάρους. Επίσης καταλαβαίνουμε, για να πω και κάτι θετικό, ότι υπάρχει από την πλευρά όλων αυτών των επιχειρήσεων αντίληψη ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Αναγνωρίζουμε ότι ήταν όλοι πρόθυμοι για να δώσουν κάποιες εξηγήσει και να επιβεβαιώσουν τη στήριξη της διαδικασίας BEPS, δηλαδή την γραμμή του ΟΣΑ. Μιλώ για την διάβρωση της βάσης και την μετατόπιση του κέρδους. Εδώ υπάρχει επί της αρχής συμφωνία και για την CCTV όταν μιλάμε για τη δημιουργία δηλαδή μιας προλογικής βάσης, τον υπολογισμό του εισοδήματος πρέπει να φορολογείται, που να είναι κοινή για όλους. Να υπάρχει συγκρισιμότητα έστω των φορολογικών συντελεστών, των φόρων, των μορφικών φόρων στις διάφορες χώρες. Και επίσης καταγράφουμε ότι υπάρχει προθυμία, επί της αρχής τουλάχιστον, να γίνεται υποβολή εκθέσεων αναχώρα, όπως πολλές επιχειρήσεις έθεσαν ανησυχίες για την δημόσια προβολή των εκθέσεων αυτών Δεν ζητούμε πλήρη διαφάνεια βεβαίω, απλώς τις βασικές πληροφορίες σε κάθε περίπτωση. Ε, επιπλέον επιβεβαιώνεται η δυνατότητα, η ανάγκη μάλλον, να έχουμε κοινή αντίληψη και αναγνωσή του τι αποτελεί φορολογική ποια χώρα είναι φορολογικό παράδεισο. Να έχουμε μια κοινή πολιτική που να επιτρέπει να αποφεύγουμε αυτέ τι μαύρε τρύπε στο σύστημα τη διεθνού φορολογία. Ω προ την διαφάνεια των φορολογικών ε, συμφωνιών σε επίπεδο εθνικό δεν δημιουργεί προβλήματα. Απλώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση που ανέφερε και η Google. Ότι εμείς είμαστε αυτοί που κάνουμε και σχεδιάζουμε την νομοθεσία. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη να συνεχίσουμε και θα δούμε τι συνέχιση πρέπει να δώσουμε στο έργο της Επιτροπής μας από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Είμαστε πάντως διαθέσιμοι για να συνεχίσουμε τον επικοδομητικό διάλογο ώστε οι πολίτες να αισθανθούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη φορολογία, στο φορολογικό σύστημα και οι επιχειρήσεις να αλλάξουν σε κάποιο βαθμό τις πρακτικές τους, διότι αυτές που τώρα χρησιμοποιούν δεν λειτουργούν και αρχίζουν να γίνονται κάποιες καταστάσεις μη βιώσιμες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Λίζα. Ο Μιχαήλ Τόιρες. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω ότι είναι σωστό αλλά και απαραίτητο ε, να κάνουμε τη σημερινή ακρόαση. Επιβεβαιωθήκαμε και διαρωτώμε για ποιο λόγο οι εκπρόσωποι των εταιριών δεν δέησαν να έρθουν πολύ νωρίτερα. Η συζήτηση είναι πολύ επικοδομητική σήμερα και πάρα πολύ νυφάλια και έδειξε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίρνει σοβαρά το ρόλο του. Και δεν υπάρχει λόγος να μην έρχονται οι εκπρόσωποι των πολυεθνικών στο Κοινοβούλιο. Και προσβλέπω σε συνέχιση ε, αυτής της προσπάθειας, αν έχουμε και περισσότερο χρόνο παράταση δηλαδή των εργασιών μας, θα ήθελα να το ξαναπούμε. Και θέλω να τονίσω ότι ορισμένα σημεία χρειάζονται περαιτέρω διευκρίνηση, τουλάχιστον σε μένα αυτό ε, σημειώνω ότι εκπρόσωποι πολλών εταιριών είπαν ότι από τη μια αξιοποιούν μόνο τις νόμιμες δυνατότητες βελτιστοποίησης φορολογίας και μάλιστα δεν έχουν μόνο το δικαίωμα αλλά καμιά φορά και το καθήκον ε, ε, των ε, μάνατζερ απέναντι στους μετόχους. Επίσης σημειώνω αυτά που είπαν οι πρόσωποι της Google και της Facebook αλλά και άλλων. Οι δύο το είπαν ξεκάθαρα αυτό ότι θεωρούν ότι με κάποιες κατασκευές και με τη διεύθυνση IP από τη, τα νησιά Καϊμάνη, από τις Βερμούδες, δεν θα πρέπει να προκύψει μειονέκτημα για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τους φορολογουμένους, αλλά μόνο για τις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Ισχύει κάτι τέτοιο και με αυτή την ε, γενίκευση. Ε, μήπως υπάρχουν αρνητικές συνέπειες γενικότερα. Γιατί αυτά τα γενικά ε, που λέμε ότι τα έχουμε στις καλένδες και θα γίνουν του Αγίου ποτέ ή το 2300 ξέρω όπως είπε ο πρόεδρος ηρωνικά και μέχρι τότε το, να υπάρχουν τέτοιες χρηματικές ροές αφορολόγητες και να χρησιμοποιούνται για να βελτιστοποιηθούν τα κέρδη και να μεγιστοποιηθούν και αυτό να είναι εις βάρος κάποιων ε, ε, Ανταγωνιστικό μειονέκτημα δηλαδή. Άλλο που θέλω να υπογραμμίσω. Ακούστηκε ένα επιχείρημα ε, που έχει να κάνει με την αμοιβαιότητα. Δηλαδή, συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στη δική μας έκθεση Έχουμε αντίστοιχη ρύθμιση, μάλλον διατύπωση ή σύσταση, ότι στις διαπραγματεύσεις και στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία για όλα αυτά τα θέματα. Τουλάχιστον αυτό να φιλοδοξούμε. Βεβαίως όλα αυτά για να γίνουν ε, θα πρέπει να ειδωθούν από κοινού με τις συστάσεις ε, του ΩΣΑ για τα BEPS. Βέβαια όλα αυτά είναι soft law, δηλαδή είναι ήπιο δίκαιο, κάπως θελοντικό και πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε υποχρεωτικό και δεσμευτικές συμφωνίες. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να μπει σε μια νομοθεσία πλαίσιο που να είναι δεσμευτική στο εσωτερικό της. Και αυτό είναι και ένα ισχυρό επιχείρημα απέναντι στις ΗΠΑ. Γιατί εάν δεν εφαρμοστεί και στην Αμερική, ε, αυτό είναι μειονέκτημα για τις εταιρείε ανταγωνιστικό, οπότε θα πρέπει να πιέσουν και με τα λόμπι να αναγκάσουν και τις Ηνωμένε Πολιτείε να το εφαρμόσουν. Και κάτι άλλο που κάπως διαφάνηκε ε, είναι η ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια και για κοινή διαχείριση ε, και αντιμετώπιση αυτών των λεγόμενων φορολογικών παραδείσων από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Φάνηκε ότι πολλές, χώρες, πολλές εταιρείες είναι παρούσες εκεί για λόγους παραδοσιακούς από ό,τι ακούσαμε, ιστορικούς, ξέρω εγώ, παραμένουν. Καλά, οι παραδόσεις αλλάζουν και αυτές, δεν είναι υποχρεωτικές. Αν δεν υπάρχουν ουσιαστικά πλεονεκτήματα να είσαι κάπου, να έχεις μια παρουσία, για ποιο λόγο θα πρέπει να διατηρήσει, ε, είναι μόνο για ιστορικούς και παραδοσιακούς μου φαίνεται λίγο αξιόπιστο αυτό το επιχείρημα, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Όχι ότι είμαστε από παλιά και τώρα που να σηκωνόμαστε να φεύγουμε. Θα πρέπει να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα έχουμε προτάσεις στην έκθεσή μας. Συνοψίζω. Κόμμα. Μάθαμε χρήσιμα πράγματα, κάποια ερωτήματα άλλα παραμένουν εκκρεμή. Ε, κατά την άποψή μου δεν έχει λυθεί ικανοποιητικά τι γίνεται με τις ρυθμίσεις ε, στο Λουξεμβούργο, στις κάτω χώρες ή στην Ιρλανδία. Γιατί υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες, ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Ποιος το ξεκίνησε αυτό, οι εκεί κυβερνήσεις, ποιος έκανε αυτή την πρόταση, ε, με αυτή την επιθετική πήγανε και στρατολογούσαν εταιρείε, δηλαδή οι κάποιοι σύμβουλοι, το management μια εταιρεία, ποιο το άρχισε αυτό, ποιο ήρξε το χειρόν αδίκο. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αυτό να το διερευνήσουμε και να το ε, ε, ε σαφηνίσουμε. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ ε, και τα μέλη του πάνελ και τους εισηγητές και τα μέλη της Επιτροπής μας όλους. Λοιπόν, τι ακούσαμε. Αυτά που ακούσαμε επιβεβαιώνουν ότι είμαστε πραγματικά σε μία καμπή και αλλάζουμε πραγματικά ρότα. Βεβαίως και, και θα χρειαστεί χρόνο. Ε, είναι κάτι το αναπόφευκτο και ακαταμάχητο. Το είπε και η Ελίζα Φεραίρα. Οι εταιρείε εδώ και 20 περίπου χρόνια έχουν καταλάβει ότι εκτός από το ουσιαστικό και θεμελιώδη οικονομικό τους ρόλο έχουν και μια κοινωνική ευθύνη απέναντι στους εργαζομένους, τους καταναλωτές και πιο πρόσφατα κατάλαβαν οι εταιρείε ότι είχαν και μια ευθύνη περιβαλλοντική, παρακαλώ. Ξέρετε ότι προετοιμάζουμε τώρα την διάσκεψη των Παρισίων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Και οι περισσότερες από τις δικές εταιρείε έχουν συνεισφέρει και στην ίδια τους τη διαφήμιση προβάλλουν ότι είναι καλοί μαθητές του περιβάλλοντος για την προστασία κτλ. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο τώρα υπάρχει και μια τρίτη διάσταση που θα πρέπει ε, και μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα καλό επιχείρημα πολίσεων είναι ότι έχουμε και ε, μια ε, ευθύνη ως πολίτες και συμμετέχουμε στη χρηματοδότηση των δημοσίων υπηρεσιών, υπηρεσιών που προσφέρονται και από τις οποίες υποφελούνται οι εργαζόμενοι σας, οι πελάτες σας, οι διευθυντές σας και όλοι μας. Αυτό το έχουν καταλάβει τελευταία κυβερνήσεις, ε, οι διοικήσεις, οι κρατικές και επίσης οι εκπρόσωποι ορισμένων πολυεθνικών. Ακόμα και αν υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά, το είπαν και οι συγητές, και πολλά σημεία που πρέπει να διευκρινιστούν και πρόοδοι να ε, επιτευχθούν. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω στα μέλη της Επιτροπής μας ότι αμέσως ε, μετά, ε, πριν τη συνεδρίαση στις 3 ε, συνεδριάζουν οι συντονιστές. Και θέλουμε να ζητήσουμε δύο πράγματα από τη διάσκεψη των προέδρων των πολιτικών ομάδων που θα συνεδριάσει την Πέμπτη. Το πρώτο είναι να μας επιβεβαιώσουν ότι η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την έκθεσή μας θα γίνει την άλλη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Στις 25 του μηνός μάλλον, το πιθανότερο, και μέχρι τότε να μπορούν να κάνουν τροπολογίες οι πολιτικές ομάδες. Και επίσης μάλλον όσο ακούσαμε σήμερα θα οδηγήσουν σε τροπολογίε από πλευράς πολιτικών ομάδων. Η δεύτερη απόφαση που λάβαμε να ζητήσουμε από τη διάσκεψη των Προέδρων παράταση εξάμηνη των εργασιών μας. Διατηρούμε λοιπόν την ημερομηνία ε, της συζήτησης για την ε, για την άλλη εβδομάδα για να μην χαλαρώσουμε από πλευρά ρυθμών. Αν θέλουμε αυτή η αλλαγή νοοτροπία να γίνει και αλλαγή νομοθεσία και αλλαγή των διεθνών συνθήκων και των φορολογικών συμβάσεων, αν θέλουμε όλα αυτά να χαραχθούν στο μάρμαρο, θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το ρυθμό. Το πρώτο έχει να κάνει με τι. Ε, αιτήσει δικαστικής συνδρομή για τα rulings και τώρα τα κείμενα που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποτελέσουν τη νομική βάση για την ενοποιημένη κοινή φορολογική βάση των εταιριών και στη συνέχεια θα πρέπει να εφαρμοστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, οι συστάσεις του ΟΣΑ. Λοιπόν, για να μην χαλαρώσουμε λοιπόν, όχι μόνο από πλευρά ρυθμού, πρέπει να ε, διατηρήσουμε και την πολιτική πίεση. Άλλος, πώς τα κράτη-μέλη που έχουν και άλλα βάσανα τώρα, δυστυχώς, αυτή την περίοδο, έχουν μεγάλες έννοιες και τραγικές πολλές φορές. Θα ψάξουν να βρουν την πρώτη δικαιολογία και την πρώτη πρόφαση για να ε, αναβάλουν κάποιες δύσκολες αποφάσεις, οι οποίες είναι σημαντικές όμως. Επαναλαμβάνω ότι επιβάλλουμε στις εταιρείες μας μικρές, μεσές και μεγάλες ένα φορολογικό σύστημα που ήταν κοπής του περασμένου αιώνα. Πριν από 100 χρόνια έχει δημιουργηθεί και δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εταιρείες ούτε στις σύγχρονες κοινωνίες. Θα πρέπει λοιπόν να να δράξουμε την ευκαιρία αυτή του σκανδάλου ή της κρίσης και δυστυχώς έτσι προοδεύουν και λειτουργούν οι δημοκρατίες για να κάνουμε τις απαραίτητες εξυγχρονιστικές προσπάθειες. Ευχαριστώ. Λύεται η συνεδρίαση. Και κανονικά είναι η τελευταία συνεδρίαση με βάση την τωρινή εντολή, αλλά βέβαια ε, εναπόκειται στη διάσκεψη των Πρόεδρων να αποφασίσει τι θα γίνει. Αν δεν παραταθεί η εντολή μας και είναι αυτή όντως η τελευταία συνεδρίαση εσχάτη, ε, σας προτείνω να συνεδριάσουμε και στο Στρασβούργο, να συναντηθούμε, να γιορτάσουμε τις εργασίες μας και τα ε, συμπεράσματα. Αν παραταθεί η λειτουργία μας βεβαίως θα τα ξαναπούμε εν ευθέτω χρόνο λήξη συνεδρία.